Καλησπέρα σε όλους. Καταρχήν, η έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Δεν βλέπω να έχει κανείς αντιρρήσεις. Μετά έγκριση των πρακτικών της συνεδρίας της 16 και 17 Δεκεμβρίου έχουν διανεμηθεί δεν βλέπω και εδώ να ακούγεται καμία αντίρρηση. Φαντάζομαι εγκρίνονται λοιπόν και τώρα με μεγάλη χαρά ερχόμαστε στον οικονομικό διάλογο και ανταλλαγή απόψεων με την Προεδρία του Συμβουλίου με τον Υπουργό Οικονομικών της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα. Ελπίζω να ακολουθηθεί η συνήθις διαδικασία, δηλαδή θα γίνει μια εισήγηση δεκάλεπτη από τον Υπουργό και μετά ερωταπαντήσεις. Ήδη έχουμε ονόματα εκείνων που ζήτησαν το λόγο σύμφωνα με τη διαδικασία των... Σημειώνω ότι οι απαντήσεις του κυρίου Στουρνάρα στους δημοσιογράφους θα, ότι θα γίνει εξ όχι μιας χώρας που πλήττεται από την κρίση αλλά εξ του Συμβουλίου. Και αναμένουμε να ακούσουμε νεότερα για τον παπάνω προϋπολογισμό και την, τις αναπτυξιακές του ρήτρες και πρωτογενές πλεόνασμα κλπ. Ξέρω ότι κι εσείς και ο Πρωθυπουργός σας είστε αισιόδοξοι ως προς τις αγορές. Με αυτό το αισιόδοξο πνεύμα λοιπόν προσμένουμε να ακούσουμε πώς θα συμπληρωθεί η νομοθεσία που πρέπει να συμπληρώσουμε τις τελευταίους αυτούς μήνες της θητείας του Κοινοβουλίου. Σας δίνω το λόγο. Thank you, Madam Chair. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μη που είμαι σήμερα μαζί σας και θα προσπαθήσω πρώτον ε, να ε, σας διαβάσω ποιες είναι οι προτεραιότητές μας ε, και κατόπιν να προσπαθήσω να απαντήσω σε ό,τι ερωτήσεις μπορεί να έχετε. So, honorable members of the committee... Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Αναλαμβάνουμε την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό αποτελεί για την Ελλάδα πραγματική πρόκληση. Αναμένεται η Προεδρία είναι δύσκολη όσο και απαιτητική, η τελευταία ε, πριν από τις ευρωεκλογέ του Μαΐου. Η οικονομική κρίση στην Ευρώπη, η ψηλή ανεργία, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων στις χώρες της Νοτιού Ευρώπης, καθώς επίσης και η κοινωνική ανασφάλεια, προκάλεσαν φωνές που αμφισβητούν ε, την κοινή μας ευρωπαϊκή πορεία. Η Ελλάδα μια χώρα που έζησε την αλληλεγγύη των Ευρωπαίων εταίρων της, καλείται τώρα να ενισχύσει και να αναδείξει όλα αυτά τα στοιχεία που μας ενώνουν. Προωθώντας έτσι περαιτέρω την ολοκληρώση, ενισχύοντας την ε, κοινωνική συνοχή, εξασφαλίζοντας την ευημερία και τη σταθερότητα για όλους τους πολίτες με την επιστροφή στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Γνωρίζουμε ότι το χρονικό μας πλαίσιο είναι περιορισμένο δεδομένου ότι η τελευταία σύνοδος ολομελίας του Κοινοβουλίου θα διεξαχθεί τον Απρίλιο. Για το λόγο αυτό και με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η Προεδρία μας ε, θα είναι de facto ε, έμπρος το βάρης. Από το 2009 η Ελλάδα ε, είχε γνωρίσει κάποια προβλήματα και σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που το αναφέρετε και υπέφερε όλες τις ε, συνέπειες και μάλιστα ήταν ε, στην καρδιά της πιο μεγάλης οικονομικής κρίσης παγκοσμίως από το 1929 χάρη στις θυσίες του ελληνικού λαού και βεβαίω στην υποστήριξη των Ευρωπαίων εταίρων μας όλα όσα ισχυρίστηκαν όσοι θεωρούσαν ότι θα βγαίναμε από την Ευρωζώνη έχουν διαψευστεί. Έχουμε ήδη κάνει δύο βασικές στρατηγικές επιλογές ως χώρα. Η πρώτη το 1981 όταν γίναμε τμήμα της ευρωπαϊκής οικογένειας που συνεχώς διευρύνεται έκτοτε. Το δεύτερο το 2001 όταν ενταχθήκαμε στον πυρήνα αυτής της οικογένειας ε, που είναι η Ευρωζώνη. Σήμερα αναλαμβάνουμε την Προεδρία, όπως είπατε, όχι ως χώρα σε κρίση, αλλά ως χώρα σε ανάκαμψη. Επιθυμούμε να συμβάλλουμε στην εμβάθυνση και στην ενίσχυση ε, της οικονομικής και πολιτικής συνεργασίας μας βασιζόμενη στα σημαντικά αποτελέσματα της Λιθουανικής Προεδρίας. Θα ήθελα τώρα να ε, ε, εξάρω τον ομόλογό μου κύριο Ριμάντα Σάτζιους που με πολύ μεγάλη αίσθηση ευθύνη κατάφερε να προωθήσει τα θέματα και μάλιστα με πάρα πολύ μεγάλη σύνεση. Είχαμε στην Αθήνα συνεδριάσεις με ε, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τη διάσκεψη των πρόεδρων του Κοινοβουλίου, καθώς επίσης και τα διάφορα πολιτικά κόμματα και πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου πριν την αρχή ακόμα της ε, Προεδρίας. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμες αυτές οι συνεδριάσεις και είχαμε την ευκαιρία να ε, ενημερωθούμε εγκαίρως και να γνωρίζουμε τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στο άτυπο συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ που θα διεξαχθεί στη ε, Αθήνα 1η και 2 Απριλίου του 2014 και σας προσκαλούμε ε, κυρία Πρόεδρε, θα επιθυμούσαμε να παρευρεθείτε. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης, τους τρόπους αντιμετώπισης τους, καθώς επίσης να εξετάσουμε και πιο αποτελεσματικούς τρόπους για τη χρηματοδότηση της οικονομίας, ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ας έρθω τώρα στην ε, Τραπεζική Ένωση. Είναι προαπαιτούμενο για περισσότερη εμπιστοσύνη και ε, οικονομική ε, αξιοπιστία, καθώς επίσης και αύξηση της ρευστότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας με διαφύλαξη της χρηματοστοπικής σταθερότητας. Ε, συμφωνούμε για τις ε, τραπεζικές εγγυήσεις και για την οδηγία για την ε, ανάπτυξη και εξυγίαση των τραπεζών και θα εξασφαλίσουμε την ομαλή ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας στην παρούσα θητεία του Κοινοβουλίου. Ο ενιαίος μηχανισμός εξυγίασης είναι εκ των όνων κάνευτής της Τραπεζικής Ένωσης, άρα πολύ μεγάλη προτεραιότητα της ελληνικής προεδρίας. Η ολοκλήρωση του μηχανισμού SRM κατά τη διάρκεια της παρούς είναι πολύ σημαντική. Συμφωνούμε όλοι ότι ο κάθε συμβιβασμό θα πρέπει να εξασφαλίζει την αποδοτικότητα, την αποφασιστικότητα, την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία του μηχανισμού. Μετά τη συμφωνία του Δεκεμβρίου για τη γενική προσέγγιση, οι τριμερεί διάλογοι έχουν αρχίσει από νωρί, ε, αρχέ Ιανουαρίου. Ε, φιλοδοξούμε να φέρουμε πιο κοντά τι θέσει Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για να επιτύχουμε μια συμφωνία που να είναι αποδεκτή από όλα τα μέρη. Έχουμε πλήρη επίγνωση ότι θα έχουμε λίγο περισσότερα στη διάθεσή μας από ένα τρίμηνο για να το ολοκληρώσουμε. Γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικός παράγωνο χρόνος και θα πρέπει να είμαστε ευέλικτοι, ε, υπεύθυνοι και να ε, τονίζουμε πάντα ότι χρειάζεται εμπιστοσύνη των πολιτών και σταθερότητα και πιο ισχυρή ευρωζώνη. Η Ελλάδα, αναλαμβάνοντας την Προεδρία του Συμβουλίου ΕΚΟΦΗΝ, θα εργαστεί προς μεγαλύτερη ευάθυνση και ολοκλήρωση της ΟΝΕ και για την ενίσχυση του συντονισμού των εθνικών οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών για να διασφαλίσουμε την ακεραιότητα του κοινού νομίσματος και να αυξηθούν οι μεταρρυθμίσεις. Στο ίδιο πλαίσιο η ελληνική προεδρία θα επικεντρωθεί στον τρόπο ενίσχυσης της κοινωνικής διάστασης της ΟΝΕ. Θεωρούμε ότι η διάσταση αυτή είναι προαπαιτούμενο για μία ε, ευρωζώνη συνεκτική και αλληλέγγυα. Πιστεύουμε ότι η εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών θα πρέπει να συνοδεύεται από πολιτικές φιλικές προς την ανάπτυξη και τις κοινωνικές πολιτικές. Αλλιώς θα οδηγήσει σε παρατεταμένη λιτότητα και θα ευνοήσει τον ευρωσκεπτικισμό. Θα ήθελα να ασχοληθώ τώρα με το, Ευρωπα... με το εξάμεινο. Ε, ήταν ιδιαίτερη ευχαρίστηση που ε, συμμετείχα στην διάσκεψη των κυβερνητών που ολοκληρώθηκε σήμερα και που ε, οι αμφιτρίονές του ήταν το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αποτέλεσε ένα ανοιχτό φόρουμ έτσι ώστε να υπάρξει ειλικρινής διάλογος και να βρεθούν τρόποι για την ενίσχυση των δημοκρατικών στοιχείων που αφορούν τη διαδικασία λήψη απόφασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα επίπεδα να ενισχύσει επίσης ε, ε, την συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού και των Εθνικών Κοινοβουλίων η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου ε, ήταν επιτυχής ε, για την ε, Ιρλανδία και επομένως είναι πολύ θετικό που πλέον αναλαμβάνει το τέταρτο εξάμεινο η Ελλάδα και ευελπιστούμε ότι θα, η επιτυχία του θα διασφαλιστεί. Έχει βάση του προγράμματος της κοινοβουλευτικής εβδομάδας αποδειχθεί ότι το πρόγραμμα είναι σωστό, ότι μπορεί να προωθηθεί η συστηματική αξιολόγηση των μεταρρυθμίσεων στην Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση, δε οι ε, ε, πολιτικέ αυτές και οι στρατηγικέ οι οποίε είχαν ήδη καθοριστεί από το Δεκέμβριο ε, στη διάρκεια του Συμβουλίου και για πρώτη φορά συμπεριλαμβάνεται και μια γενικότερη έποψη της, του, του τρόπου με τον οποίο έχουν υλοποιηθεί οι συστάσεις οι οποίε είχαν γίνει τον προηγούμενο Ιούνιο. Θεωρούμε ότι και τα οικονομικά και τα κοινωνικά στοιχεία λαμβάνονται σωστά υπόψη μέσω των συμβουλίων ε, ΕΚΟΦΗΝ και ΕΝΚΟ ε, και αυτό στη διάρκεια του επόμενου εξαμήνου. Επίσης, ε, θα ε, υπάρχει η πρόθεση από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, να υπάρξουν συγκεκριμένες συστάσεις και εκθέσεις ανά χώρα έτσι ώστε να γίνει σεβαστό το χρονοδιάγραμμα. Οι μακροοικονομικές ανισορροπίες έχουν γίνει σημαντικό στοιχείο έτσι ώστε να υπάρξει βελτίωση της οικονομικής εικόνας. Ορισμένες συστάσεις του Ιουνίου βασίζονται ακριβώς σε αυτή τη διαδικασία. Ιδιαίτερη προσοχή ε, θα δοθεί στις συστάσεις αυτές στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η μακροοικονομική ε, ε, ε, εικόνα της οικονομίας. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν 99% των επιχειρήσεων και 17% των θέσεων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται λοιπόν για ένα κυρίαρχο στοιχείο για την οικονομική ανάκαμψη. Αυτό το αναγνωρίζει η Ελληνική Προεδρία και επομένως ε, θέλει να διευκολύνει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς επίσης μέσω αυτών να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Θεωρούμε ότι ιδιαίτερη σημασία ε, έχουν ε, πολλές προτεραιότητες, όπως ας πούμε η κοινή πρωτοβουλία της Τράπεζας Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενδυνάμωση της οικονομίας, κυρίως δε ε, η διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, για την ε, ε, αύξηση κεφαλαίου των επενδύσεων καθώς επίσης και την χρηματοδότηση των προγραμμάτων υποδομών που αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η έλλειψη ρευστότητας οπωσδήποτε ήταν πάρα πολύ σημαντική και επιδίνωσε την κρίση. Μέχρι τώρα δε έχει υποβαθμιστεί κυρίως όσον αφορά τις οικονομίες των περιφερειακών χωρών της Ευρώπης που βρίσκονται ε, σε ε, ιδιαίτερη οικονομική δυσκολία. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, οι απαραίτητες δράσεις έτσι ώστε να σταματήσουν η φοροαποφυγή και η φοροδιαφυγή στοιχεία τα οποία επιβαρύνουν την οικονομική κατάσταση των χωρών. Η Ελληνική Προεδρία με μεγάλη προσοχή θα παρακολουθήσει την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων με τρίτες χώρες περιλαμβανομένης και της Ελβετίας ε, ε, σύμφωνα και με την ε, σύσταση η οποία, και την εντολή η οποία έγινε ε, η οποία της εδόθη τον, ε, την άνοιξη του 2013. Επίσης ε, θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε έτσι ώστε να υπάρχει αυτόματη ανταλλαγή φορολογικών στοιχείων μεταξύ των κρατών μελών αλλά και μεταξύ τρίτων χωρών και χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να παρέχει συντονισμένο input στην ήδη σοβαρή δουλειά του ΟΑΣΑ καθώς επίσης και με γενίκευση του συστήματος ανταλλαγής στοιχείων και πληροφοριών. Ε, τη στιγμή που τα δημόσια οικονομικά πιέζονται πάρα πολύ σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστεύουμε ότι θα πρέπει ε, οπωσδήποτε ε, οι φορολογικές βάσεις να μην διαβρωθούν περαιτέρω. Το Συμβούλιο ε, προσπαθεί να ε, δει το θέμα αυτό και μέσω της ε, οδηγίας για την επικουρικότητα. Όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, γνωρίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί το Κοινοβούλιο και το στηρίζει το Κοινοβούλιο. Θα συνεχίσει η Ελληνική Προεδρία τους επόμενους μήνες να ασχολείται με το θέμα η Πολυθωνική Προεδρία φτάσαμε στην ολοκλήρωση ενός πρώτου τμήματος τώρα. Ε, θα πρέπει η Πολυνική Προεδρία να ε, αποσαφινιστούν κάποια στοιχεία, ε, κάποια τεχνικά, κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν την ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Θα ήθελα τώρα να ασχοληθώ με ένα άλλο θέμα που είναι η αναθεώρηση της εποπτικής αρχής το, ε, ε, η εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα είναι κάτι που μας απασχολεί πάρα πολύ ε, και ε, θεωρούμε ότι η αναθεώρηση θα πρέπει αυτής θα οδηγήσει σε αύξηση της ρευστότητας. Είναι ένα θέμα το οποίο γνωρίζουμε ότι απασχολεί το Κοινοβούλιο και σχετίζεται βεβαίως και με την μύφλα. Είναι ένα σημαντικό βήμα έτσι ώστε να έχουμε υγιέστερο, πιο διαφανές αλλά και πιο υπεύθυνο ε, ε, και υγιές ε, οικονομικό σύστημα. Με τους αναθεωρημένους κανόνες θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα την κρίση και επομένως να μειωθούν οι συστημικοί κίνδυνοι. Ταυτοχρόνως δε να διασφαλιστεί η σταθερότητα των χρηματαγορών. Όσον αφορά την οδηγία, την πρόταση οδηγίας για το benchmarking, καταλαβαίνω κυρία Πρόεδρε ότι είστε ε, εισηγήτρια για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Σε αυτόν τον ε, τομέα θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε την εργασία στο Συμβούλιο όσο γίνεται περισσότερο. Συμφωνώ μαζί σας ότι είναι ύψιστη σημασία ε, να παραχθεί ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας και για τους καταναλωτές και για τους επενδυτές. Following Όσον αφορά τα πρίψη και ξέρω ότι συζητήθηκε το θέμα στην 20 η Νοεμβρίου ε, στο Κοινοβούλιο έλαβα ε, ε, μια επιστολή από την κυρία Μπέρεσε και της απήντησα ότι κατανοώ απολύτως την ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας των παρεχομένων στους καταναλωτές πληροφοριών και βεβαίως συμφωνώ μαζί σας ότι θα πρέπει να προωθηθεί αυτή η πρόταση. Ε, όσον αφορά την ε, ε, οδηγία την, που σας απασχολεί επίσης, όσον αφορά την ανταλλαγή στοιχείων, την 7η Ιανουαρίου συζητήθηκε το θέμα αυτό. έχει ξεκινήσει ξεκινήσει τριμερή διάλογο, και είμαι πεπισμένο ότι παρότι δεν έχουμε ήδη κοινέ θέσεις ε, θα οδηγηθούμε σε κάποια ε, συμφωνία όσον αφορά την προστασία των ε, καταθέσεων. Επίσης ε, θα προωθήσουμε ένα πιο ε, ε, ισχυρό και καλύτερα ελεγχόμενο σύστημα για τις αγορές και για τις πληρωμές έτσι ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την προστασία των καταναλωτών. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα των λογαριασμών, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η προστασία των μικρών τραπεζών επίσης θέλουμε ε, ή ε, θέλουμε το θέμα των, ε, του κόστους και των τελών που εφαρμόζουν οι διάφορες τράπεζες να ομοιογενοποιηθεί και εν πάση περιπτώσει να γνωρίζουν οι καταναλωτές μας, να γνωρίζουν οι πολίτες της Ευρώπης τι ακριβώς πληρώνουν και τι ακριβώς τους χρεώνουν. Αυτά είναι θέματα σημαντικά για την ελληνική προεδρία. Θεωρούμε ότι με τον τρόπο αυτό και θα είναι καλύτερος ο ανταγωνισμός όσον αφορά τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αλλά και θα βελτιωθεί βελτιωθεί και κοινωνικά και οικονομικά η θέση των ε, ε, πολιτών. Κυρία Πρόεδρε, γεννήθηκα σε μια χώρα η οποία αναγνωρίζει την σημασία του Κοινοβουλίου, ε, την σημασία της δημοκρατίας και βεβαίως την σημασία της ύπαρξης κοινών προτύπων τα οποία προωθούνται μέσω δημοκρατικών διαδικασιών. Θα χρειαζόμαστε λοιπόν και το Ελληνικό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι ώστε να μπορέσουμε να προωθήσουμε και να υλοποιήσουμε τις προτάσεις μας. Βασίζομαι λοιπόν στην προσπάθεια την κοινή που θα κάνουμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρο. Περνάμε <coughs> τώρα στις ερωταπαντήσεις. Έχουμε λιγάκι ξεπεράσει το χρόνο μας ήδη. Παρακαλώ λοιπόν να συντομεύουν όλοι γιατί αλλιώς θα χρειαστεί να αφαιρέσω το λόγο από ορισμένους προς το τέλος. Για τους πρώτους δύο ίσως να είμαι πιο μαλακιά. Πρώτα απ' όλα λοιπόν για το ΕΛΚ. Η Κορίν Βόρτμαν Κόλ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να σας ευχαριστήσω κύριε Προεδρεύον και να σας συγχαρώ εσάς και την κυβέρνησή σας για τις προόδους που έχετε κάνει παρόλο που είναι ακόμα έφραυστα τα στοιχεία. Κάνατε τις μεταρρυθμίσεις, εξηγιάνατε τα οικονομικά σας και τώρα αρχίζει αυτό να αποδίδει. Θα ήθελα να σας ενθαρρύνω να διατηρήσετε αυτή τη φιλοδοξία γιατί αν θέλετε πραγματικά να επιταχύνετε στην οικονομική ανάκαμψη και ανάπτυξη να κατεπολεμήσετε την ανεργία χρειάζεται χρειάζεται πραγματικά φιλοδοξία. Στο ίδιο επίπεδο φιλοδοξίας όμως χρειαζόμαστε και ε, ε, να αντιμετωπίσουμε τα ευρωπαϊκά ζητήματα με την ίδια φιλοδοξία για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης. Και πραγματικά μας λυπεί το γεγονός ότι όταν ε, βλέπει κανείς τη θέση του Συμβουλίου. Αυτό που από κοινού αποφασίσαμε και προτείναμε ήταν ένας ουσιαστικά ενιαίος μηχανισμός για την εξυγίανση. Ε, η θέση του Συμβουλίου πρέπει να πω ότι μας ανησυχεί βαθύτατα, δεν βοηθάει στην επίτευξη του στόχου. Να σας δώσω τρεις βασικούς λόγους που το λέω αυτό. Το σύστημα διακυβέρνησης που προτείνει το Συμβούλιο είναι πάρα πολύ περίπλοκο δεν μπορεί μια τράπεζα να εκαθαριστεί μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Χρειαζόμαστε ένα ταμείο με ε, ίδια μεταχείριση των τραπεζών ανεξαρτήτως του κράτους μέλους το οποίο εδρεύουν. Η κατάσταση λοιπόν είναι ε, πάρα πολύ σοβαρή, πάρα πολύ κρίσιμη και πρέπει να συμφωνήσουμε οπωσδήποτε πριν από τις ευρωεκλογέ. Αυτό όμως τι σημαίνει, ότι θα πρέπει να έχετε και φιλόδοξη εντολή. Το επίπεδο της εντολής δεν ανταποκρίνεται ε, στη θέση του Συμβουλίου. Όταν λάβετε την εντολή αυτή, ξέρετε πότε θα είναι, γιατί τότε θα αρχίσουμε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. Και δεύτερον, δεν συμφωνούμε με μια διακυβερνητική συμφωνία. Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να είναι συμπληρωματική προς τον κανονισμό αυτή. Μπορείτε να μας επιβεβαιώσετε αυτό που μας υποσχέθηκε ε, το Συμβούλιο στον Τριμερή Διάλογο ότι η ε, κυβερνητική ε, συμφωνία δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί πριν καταλήξουμε εμείς για το μηχανισμό εξηγίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Πράγματι, στην Ελλάδα έχουμε υψηλές προσδοκίες και φιλοδοξίες και έχουμε ήδη πετύχει τους περισσότερους στόχους από τους, τους οποίους είχαμε θέσει για την αρχή και για την ανταγωνιστικότητα και για τα δημοσιονομικά τώρα. Για την Τραπεζική Ένωση. Όλοι συμφωνούμε ότι θέλουμε μια ισχυρή Τραπεζική Ένωση γιατί πήραμε μαθήματα από την κρίση. Συμφωνούμε λοιπόν πλήρως για την έννοια του steady state. Τώρα μπορεί να διαφέρουμε στις μεθόδους. Στο Συμβούλιο πολλούς μήνες συζητήθηκαν οι μεθοδολογίες και νομίζω ότι επιλέξαμε την λιγότερο επικίνδυνη οδό. Καταλαβαίνω βέβαια ότι θα υπάρξουν διαφωνίες. Χρειάζεται πιο πολύ αμοιβαία κατανόηση για τη διαδικασία. Γιατί όπως είπε και ο Καβάφης, δεν είναι σημαντικό μόνο ο προορισμός να φτάσουμε στην Ιθάκη, αλλά και το ταξίδι το ίδιο είναι σημαντικό. Εμείς ως Ελληνική Προεδρία θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη κατανόηση της κατάστασης. Ας μην υπησέλθω σε λεπτομέρειες. Οι διαπραγματευτές θα το κάνουν αυτό για να επιτευχθεί ο κοινός στόχος. Συμμεριζόμαστε όμως την άποψη ότι είναι απολύτως ζωτικό να υπάρξει συμφωνία τελικά. Γιατί μια ευρωζώνη χωρίς μια ισχυρή τραπεζική ένωση θα, δεν θα ήταν πλήρης. Ε, θέλω να ρωτήσω συμπληρωματικά κάτι. Μπορείτε να μας επιβεβαιώσετε ότι το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ δεν θα καταλήξει σε διακυβερνητική συμφωνία πριν να έχει βρεθεί συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για την Τραπεζική Ένωση. Δεν μπορώ να το βεβαιώσω. Δεν μπορώ να βεβαιώσω γιατί πρέπει πρώτα να το συζητήσω με τους συναδέλφους μου στο Συμβούλιο. Okay, well, it'll all come back to bite you. Καλά. Θα επανέλθουμε να σας δαγκώσουμε αν ε, κάνετε κάτι τέτοιο. Ελίσα Φερέρα. Θα ξεκινήσω από εκεί που σταμάτησε η συνάδελφος ε, Φόρτμαν. Καταλαβαίνετε ότι το Κοινοβούλιο είναι ενωμένο εδώ. Έτσι. Έχουμε βεβαίως ε, συγκεκριμένη θέση την οποία έχουμε υπερψηφίσει κατά 80%. Το τελευταίο σας ε, σχόλιο μας εκπλήσει και είναι σοβαρή η έκπληξή μας γιατί είχαμε την εντύπωση ότι η διακυβερνητική συμφωνία, βάσει του τριμερούς διαλόγου δηλαδή, δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί πριν εμείς ολοκληρώσουμε τις συμφωνίες για το SRM καταλαβαίνετε ότι εμείς αμφισβητούμε κατά κάποιο τρόπο την νομιμότητα της διαδικασίας εάν δεν προχωρήσει με τον τρόπο αυτό ε, και επομένως ε, ε, γνωρίζομαι ότι θα πρέπει να συνεχίσει η διαδικασία και σύμφωνα με την ευχή του Κοινοβουλίου θα πρέπει να γίνει ένας πρώτος έλεγχος. Κοιτάξτε, αναφέρατε ότι θέλετε να υπάρξει μια συμφωνία. Το Κοινοβούλιο θέλει και αυτό να έχει συμφωνία, αλλά όχι οποιαδήποτε συμφωνία. Εμείς επιθυμούμε σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια καλή συμφωνία. Είναι προφανές ότι εάν ολοκληρωθεί αυτή η εντολή, αυτή η θητεία του Κοινοβουλίου, ε, θέλουμε να έχουμε ένα σύστημα ε, για την ε, λύση των τραπεζών και την εξυγίαση των τραπεζών που να είναι σύμφωνα και με τις αρχές που έχουμε πρεσβεύσει μέχρι τώρα. Γιατί καταλαβαίνετε ότι πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει υπάρχει και μια συνέχεια, ένα follow-up το οποίο είναι οργανωμένο. Είχαμε έκοφιν στις 27, στις 28 υπάρχει και μια διακυβερνητική, αργότερα έχουμε και τριμερή διάλογο. Ε, μπορούμε να προσδοκούμε ότι τουλάχιστον κάποια στοιχεία από τις ε, θέσεις του Συμβουλίου αφήνουν κάποιο περιθώριο ελιγμών για το Κοινοβούλιο. Ε, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω δεν υπάρχει περαιτέρω εντολή για το Κοινοβούλιο, συγγνώμη, δεν υπάρχει εντολή για την ελληνική Προεδρία έτσι ώστε από μόνη της να προχωρήσει. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω, εάν εννοούμε αυτά που λέμε, τότε θα πρέπει να γεφυρωθούν με κάποιο τρόπο οι διαφορές. Δεν μπορούμε να έχουμε απέναντί μας ένα ε, συμβούλιο με παγιωμένες θέσεις που να μην έχει καμία δυνατότητα τροποποίησης. Ευχαριστώ. Απάντηση. Όπως γνωρίζετε, η διακυβερνητική συμφωνία δεν γίνεται υπό το ΕΚΟΦΗΝ. Οι Έλληνες διαπραγματευτές βεβαίως έχουν την απαραίτητη εντολή έτσι ώστε να διαπραγματευτούν μαζί σας και να βρουν λύσεις. Σε αυτή τη φάση ωστόσο δεν μπορώ να επαληθεύσω με τα βεβαιότητος ότι μπορώ να απαντήσω θετικά στην ερώτηση που ε, υποβάλατε. Ας αφήσουμε λίγο χρόνο, ας είμαστε λίγο ευέλικτοι, ας αφήσουμε χώρο ε, για τις ε, ε, συμβιβαστικές λύσεις, γιατί νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε συμβιβασμούς. Εν τέλει, αυτό που επιθυμούμε και οι δύο είναι να έχουμε μία νομική βάση η οποία να είναι ισχυρή. Επομένως, ας έχουμε μια αμοιβαία κατανόηση ας συζητήσουμε με καλό πνεύμα και με ικανό βαθμό ευελιξίας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βρούμε κοινού τόπους. Ας μην προδικάσουμε οτιδήποτε, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον. Well, I, I uh, must Πρέπει να πω ότι ε, ακούμε μια-δυο καλές φράσεις, ε, εντάξει δεν προ καταλαμβάνετε τίποτα, θέλετε να είστε βέλεκτος αυτά είναι τα θετικά. Μακάρι να τα πείτε και στο ΕΚΟΦΗΝ έτσι και να τους εξηγήσετε ε, όταν φτάσετε μια θέση που είναι στα μισά περίπου του δρόμου τα που μας χωρίζει και όχι 99% προς την κατεύθυνση του Συμβουλίου. Γιατί αυτό μάλλον δεν θα μπορέσουμε να το ανεχθούμε. Τώρα, εξ ονόματος των φιλελευθέρων, ο κύριος Βολφ Κλίντς. Κύριε Υπουργέ, Κύριε Υπουργέ, έχει πετύχει πάρα πολλά για τη χώρα σας και αυτό είναι καλό και για την Ελλάδα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και πραγματικά σας συγχαίρω ειλικρινά. Οι θετικές αυτές εξελίξεις όμως ε, για να αποδειχθούν βιώσιμες δεν αρκεί ε, και μόνο άπαξ να έχετε ε, πρωτογενές πλεόνασμα, πρέπει να δημιουργήσετε εκείνες τις συνθήκες πλαίσιο στη χώρα σας που θα προσελκύσουν πιθανούς επενδυτές. Να είστε ενδιαφέροντες ε, για να πούνε χώροι αλλά και αλλοδαποί επενδυτές, μάλιστα θα έρθουμε να επενδύσουμε. Αυτές λοιπόν οι ε, διαδικασίες και το πλαίσιο δεν υπάρχουν ακόμα και μου λείπουν. Ε, μιλώ με οικονομικούς παράγοντες από τη χώρα σας που καταγγέλουν την γραφειοκρατία που είναι ακόμα ισχυρή, πολύ βραδία η λήψη των αποφάσεων και για τις χρήσιμες πληρωμές, για να το πω έτσι, ε, είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν κάτι για να προωθηθούν τα θέματά τους στους αρμοδίους. Ε, εσείς αυτό το τομέα ε, τι σκοπεύετε να κάνετε, θα δημιουργήσετε ε, τις προϋποθέσεις για να καταπολεμηθεί ε, η ευνοιοκρατία, ο νεποτισμός και η γραφειοκρατία και η διαφθορά. Well, thank you. Ευχαριστώ κύριε Κλίντ. Θα απαντήσω ως Έλληνας Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του ΕΚΟΦΗ. Μερικές φορές λένε ότι η Ελλάδα έκανε αρκετά δημοσιονομικά αλλά όχι δομικά. Αυτό δεν είναι σωστό. Αν διαβάσετε τις εκθέσεις του ΩΣΑ για την ανάπτυξη του περασμένου χρόνου, λένε ότι από την αρχή της κρίσης η Ελλάδα ήταν πρωταθλητής στις δομικές μεταρρυθμίσεις. Πράγματι, υπάρχουν ακόμη μερικά πράγματα που πρέπει να ολοκληρωθούν δηλαδή η απελευθέρωση περισσότερων επαγγελμάτων και αγορών προς όφελος μεγαλύτερο του καταναλωτή, ε, απασχόληση, αλλά συμπληρώσαμε περίπου 70% των δομικών μεταρρυθμίσεων που απαιτούνταν και αυτό φαίνεται από την τεράστια μείωση στο κόστος της εργασίας κατά 25 περίπου της η Ελλάδα λοιπόν έχει επανέλθει στην ανταγωνιστικότητα που είχε χάσει από τότε που μπήκε στο ευρώ και ιδιαίτερα μετά το 2009. Σε τέσσερα χρόνια καταφέραμε να επαναφέρουμε την ανταγωνιστικότητα εκεί που ήταν όταν μπαίναμε στο ευρώ. Και η πρόσβαση των επενδυτών ε, κατέστη ευκολότερη. Περικόψαμε γραφειοκρατικές διαδικασίες και αντί για τη γραφειοκρατία τώρα τους ξετυλίγουμε κόκκινο χαλί τους επενδυτές. Αυτό ακόμα πρέπει να ολοκληρωθεί βέβαια. Μειώσαμε όμως τη γραφειοκρατία. Καταρχήν το μέγεθος του δημόσιου τομέα τρομερά. 200.000 λιγότεροι δημόσιοι υπάλληλοι από ό,τι το 9. Από όλε τι απόψει λοιπόν μειώσαμε το κράτος, είναι πιο αποτελεσματικό. Αδέχομαι ότι πρέπει να γίνουν κι άλλα. Αυτό μου αρέσει που είπατε. Red carpet αντί για red tape. Δηλαδή ξετυλίγουμε κόκκινο χαλί αντί για γραφειοκρατία. Αυτό μου αρέσει. Ε, αλλά θα πρέπει να, γίνει, να, να γεμίσει και σαν έννοια βέβαια. Ε. Ashley Fox. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ για την παρουσίασή σας. Η χώρα σας πήρε πολλά χρήματα για τη διάσωση το 2010 και ένα δεύτερο bailout το 2012. 110 δις την πρώτη φορά και 140 τη δεύτερη. 1,5 εκατομμύριο είναι οι άνεργοι στην Ελλάδα, 28% και 57% είναι η ενεργεία για τους νέους. Αυτό είναι εκπληκτικό. Μπορείτε να μας εξηγήσετε λοιπόν πώς βλέπετε αυτή την κατάσταση ως οικονομική επιτυχία. Thank you, Mr. Fox. I Απάντηση. Θα απαντήσω και εδώ ως Έλλην Υπουργός Οικονομικών. Δυστυχώς ε, τα οικονομικά δεν είναι άσπρα μαύρα, δεν είναι όπως η φυσική και η χημεία. Μερικές φορές ε, τα, χρονικά περιθώρια πρέπει να είναι πιο μεγάλα. Χρειαζόμαστε χρόνο. Σας είπα ότι τα αριθμητικά στοιχεία έχουν βελτιωθεί. Σας είπα επίσης ε, ότι τώρα έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα στη θέση του χαόδους ελλείμματος και στο ισοζύγιο πληρωμών επίσης η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη. Αλλά ξέρετε, ότι στα οικονομικά υπάρχει μία διάσταση χρονική ανάμεσα από τη στιγμή που τα οικονομικά νούμερα βελτιώνονται και τη στιγμή που ο κόσμος αρχίζει και αισθάνεται την αλλαγή αυτή. Επομένως, εδώ ακριβώς χρειαζόμαστε την αρρωγή των κοινωνικών εταίρων, την αρρωγή και τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έτσι ώστε να κατανοήσουν ότι έχουμε μπει στο σωστό δρόμο, να κατανοήσουν επίσης ότι στα οικονομικά δεν βελτιώνονται τα στοιχεία μέσα σε μια νύχτα, να κατανοήσουν ότι έχουμε διανύσει το 80% του δρόμου που θα μας οδηγήσει στην ολική διάσωση και να ζητήσουμε λοιπόν ε, υπομονή για αυτή τη μικρή απόσταση που υπολείπεται η κατάσταση βελτιώνεται και μάλιστα με ταχύ βήμα. Η ανεργία έχει πέσει. Λίγο, το δέχομαι. Ωστόσο έχει πέσει. Σε εννέα βιομηχανικούς τομείς έχουμε δει αύξηση των θέσεων εργασίας το τελευταίο τρίμηνο. Επομένως, έχει ξεκινήσει αυτή η θετική πορεία. Μακάρι να μπορούσα να σας φέρω ακόμα καλύτερα νέα. Όμως είμαι βέβαιος ότι όταν θα ξαναέρθω στο τέλος της ελληνικής προεδρίας θα έχω καλύτερα στοιχεία να σας δώσω, καλύτερα νέα για την ανάπτυξη ε, και για την ανεργία. Μετά από πέντε χρόνια, ενδεχομένως φέτος θα είναι η πρώτη χρονιά, είναι πολύ πιθανό αυτό, που θα έχουμε θετικό πρόσημο στην ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Βεβαίως η κατάσταση είναι ενδιαφέρουσα στην Ελλάδα. Αλλά πρέπει να σας υπενθυμίσω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι εδώ ε, θέλουμε να ανταλλάξουμε απόψεις ε, όσον αφορά τη δικιά μας τη δουλειά, τα ευρωπαϊκά. Ο ε, συνάδελφος κύριος Λάμπερτς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι δύσκολο να αντισταθεί κανείς στον πειρασμό να μιλήσει κανείς για αυτή τη μικρή χώρα που έπαιξε τόσο μεγάλο ρόλο στην ευρωπαϊκή ιστορία και στην πιο πρόσφατη. Κύριε Στουνάρα είπατε ότι δεν είναι κβαντική φυσική ε, η οικονομία μπορεί να μην είστε φυσικός, αλλά ξέρετε ότι η κβαντική φυσική είναι ένα τμήμα της ε, φυσικής που δεν είναι τόσο δετερμινιστικό. Εν πάση περιπτώσει, επειδή είμαι μηχανικός τα λέω όλα αυτά, αλλά οι οικονομολόγοι μας λένε συνεχώς ε, ότι τα οικονομικά δεν είναι ε, μια θετική επιστήμη, ε, η ακριβής επιστήμη, αλλά πρέπει να σας πω ότι περισσότερο από το μισό του πληθυσμού σας ε, δεν συμφωνεί με την έννοια που αποδίδεται στην επιτυχία και θέλει περισσότερο. Σας άκουσα να μιλάτε για τα φορολογικά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είναι χαρά μας πάντα να ακούμε το Συμβούλιο να λέγει ότι θέλουμε να κάνουμε μεγάλα βήματα στην φορολογία. Από μια χώρα όμως που έχει ε, ρεκόρ ε, ως προς την αποτελεσματικότητα δικαιοσύνης και συλλογής των φόρων ε, που δεν λάμπει με τις επιδόσεις της, επιτρέψτε μου λίγο να αμφιβάλλω. Ιδιαίτερα εγώ είμαι υπέρ ε, μιας περισσότερης δικαιοσύνης προς την Ελλάδα, δηλαδή να μην επιβάλλουμε λεόντιες ε, προϋποθέσεις και όρους για τη διάσωση της Ελλάδας, αλλά στα φορολογικά εκπλήσωμε όχι μόνο στην Ευρώπη από την έλλειψη πρόοδου αλλά και στην ίδια σας τη χώρα. Να φορολογήσετε τους πλουσίους στην Ελλάδα γιατί βλέπω ότι το κόμμα σας, το δικό σας και το ε, σύμμαχο κόμμα σας ε, είστε μάλλον στα ανώτερα στρώματα και διστάζετε να τους φορολογήσετε. Οποιαδήποτε πρόοδος ε, θα μας βρει σύμφωνος. Θα τα συζητήσουμε και την άλλη εβδομάδα αυτά στην Αθήνα. Ευχαριστώ πολύ. Θα απαντήσω για μία ακόμα φορά σαν ε, υπουργό Οικονομικών. Ένας ταπεινός οικονομολόγος είμαι, δεν είμαι κβαντικός φυσικός. Ό,τι μπορώ λοιπόν θα κάνω. Όσον αφορά την φορολόγηση, πρέπει να σας πω ότι στην Ελλάδα έγιναν τρομερές πρόοδοι. Περάσαμε ε, ε, ε, καινούριου φορολογικούς κώδικες και από το 2001 για πρώτη φορά έχουμε πλέον πλεόνασμα, δηλαδή έχουμε ξεπεράσει τους στόχους κατά 3% όσον αφορά την φορολόγηση και, την, και τους φόρους. Είμαστε λοιπόν οι μαθητές. Ε, έχουμε περάσει καινούρια, σύγχρονη, επικαιροποιημένη νομοθεσία και επομένως ε, έχουμε ε, φτάσει πλέον σε επίπεδα που προσπαθούμε πραγματικά να, απο, να, να χτυπήσουμε, να πατάξουμε την φοροδιαφυγή και την φοροαποφυγή. Γιατί καταλαβαίνετε ότι η εξαπάτηση δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά και ολόκληρη την Ευρώπη. Ε, έχω λίγο χρόνο ακόμα νομίζω. Τι γίνεται με την φορολογική ε, δικαιοσύνη, tax justice. ε, ε, ε το να ε, περνάει κανείς καινούριου φορολογικού κώδικες είναι ένα πράγμα. Το να υλοποιεί, να εφαρμόζει τους κώδικες αυτούς είναι ένα άλλο πράγμα. Και εδώ προκύπτει το ερώτημά μου και εδώ έχω αμφιβολία. δηλαδή ότι αυτοί που είναι χαμηλοσυνταξιούχοι και είναι αυτοί που στο, στους ώμους τους βαραίνει περισσότερο το φορολογικό βάρο. Απάντηση. Έχουμε κάνει ε, αναθεώρηση όλου του συστήματος ε, της φορολογίας. Ε, ξέρετε ότι η φοροδιαφυγή βασίζεται σε δύο άξονες, την δυνατότητα, το ενδεχόμενο να σε πιάσουν και το ενδεχόμενο να σε τιμωρήσουν. Εμείς αυτές τις δύο πιθανότητες τις έχουμε αυξήσει όσο μπορούσαμε περισσότερο. Έχουμε χρησιμοποιήσει ε, ε, και ε, νέα συστήματα και νέους υπαλλήλους σαν ελεγκτές. Έχουμε αλλάξει και το σύστημα κυρώσεων. Και επομένως δέστε λίγο ε, και πόσους έχουμε βάλει στη φυλακή, πλούσιους που βρίσκονται πλέον πίσω από τα σίδερα της φυλακής. Ο κύριος Χουντής. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σας καλωσορίζω και με την ιδιότητά σας ως Προέδρου του ΕΚΟΦΗΝ στην Επιτροπή μας. Θέλω να σας πω ότι και σήμερα ακούστηκαν, αλλά τον τελευταίο καιρό η ελληνική κυβέρνηση ακούει πολλά συγχαρητήρια για τα επιτεύγματά της. Ξέρουμε πολύ καλά βεβαίως ότι η Ελλάδα είναι στα όρια της ανθρωπιστικής κρίσης. Με τους δείχτες της ανεργίας των νέων αναφέρατε και ορισμένα σε αυτά. Θέλω να σας πω λοιπόν, η ερώτησή μου είναι πολύ συγκεκριμένη. Αυτό που είπατε πριν από λίγο, ότι σε τελική ανάλυση είσαστε ένας ταπεινός οικονομολόγος, ακούστηκε για πρώτη φορά πριν λίγες μέρες από τον κύριο Όλι Ρεν, ο οποίος κάποια στιγμή όταν στριμώχτηκε στις απαντήσεις αμφισβήτησε τις δυνατότητες της επιστήμης. Και γιατί σας το λέω αυτό. Σας το λέω γιατί θέλω να μου σχολιάσετε τη δήλωση ενός ταπεινού οικονομολόγου, όπως του κυρίου Όλιρε, που είπε ότι αν κουρεύαμε το ελληνικό χρέος την άνοιξη του 2010, τότε η κρίση θα μεταδίδεται και στις άλλες χώρες και στις ευρωπαϊκές τράπεζες. Δηλαδή, θυσιάστηκε ο ελληνικός λαός και η ελληνική οικονομία, δεν ξέρω αν τα συγχαρητήρια είναι για αυτές τις θυσίες, για να σωθούν οι ευρωπαϊκές τράπεζες. Και ένα δεύτερο, πιο συγκεκριμένο ερώτημα που έχει σχέση με τις προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας και το επίδικο θέμα της Τραπεζικής Ένωσης, της Τραπεζικής Εποπτείας. Σύμφωνα με όσα ξέρουμε, οι έλεγχοι που θα γίνουν κεντρικά από τις τράπεζες, το πλαίσιο αυτής της εποπτείας, θα ζητούν ως κατώτατο όριο κεφαλαϊκής επάρκειας για τις Ευρωπαϊκές Συστημικές Τράπεζες το 8%. Γνωρίζετε όμως κύριε Υπουργέ ότι λόγω μνημονίου, λόγω προγράμματος οικονομικής προσαρμογής για τις ελληνικές τράπεζες το όριο για το 2012-2014 είναι 9%. Πείτε μου σας παρακαλώ, εκτιμάτε ότι είναι μια δυσμενής αντιμετώπιση. Είναι μια αντιμετώπιση που μπλοκάρει τουλάχιστον 2 δισεκατομμύρια σε ένα γενικευμένο πρόβλημα ρευστότητας στην ελληνική οικονομία, καθώς οι τράπεζες δεν δανείζουν μικρές, μεγάλες επιχειρήσεις και ιδιώτες. Τι σκοπεύετε να κάνετε σε αυτό το σημείο. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι και εγώ κύριε Χουντή που είμαι εδώ σήμερα μαζί σας. Ε, πρώτον, θα ήθελα να πω ότι ο ελληνικός λαός πράγματι υπέστη σοβαρές θυσίες τα προηγούμενα χρόνια, όμως η κατάσταση τώρα έχει βελτιωθεί σημαντικά. Από το 2014 και μετά ε, όλες οι ενδείξεις είναι ότι θα έχουμε ε, έστω και σταθερότητα στην αρχή και μετά βελτίωση του εισοδήματος του κόσμου μετά από πολλά χρόνια ε, αύξηση της ανεργίας, μείωση των ε, πραγματικών μισθών. Όμως ε, θέλω να τονίσω ότι οι, Ευρωπαίοι, η Ευρωπαίοι εταίροι μας έχουν, έχει δείξει συνοχή, έχουν δείξει solidarity. Όπως ελέγχθη πριν από τον κύριο Φόξ, έχουμε πάρει συνολικό δάνειο περίπου 240 <laughs> εκατομμυρίων. Έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες αυτού του δανείου. Σήμερα το μέσο επιτόκιο που η Ελλάδα πληρώνει είναι περίπου λίγο κοντά στο 2%. Είναι, ένα, είναι, ένας αρκετά καλός, ε, είναι αρκετά καλή όρη. Ε, η αποπληρωμή έχει μεταφερθεί 30 χρόνια πίσω και σε λίγο, αφού τελειώσουμε τις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα, θα ξεκινήσει η συζήτηση για την περαιτέρω μείωση του ελληνικού χρέου, σύμφωνα με την νομική βάση που υπάρχει στην απόφαση του Eurogroup της, ε, 28 Νοεμβρίου του 2012 με βάση αυτή την ε, ε, νομική βάση οι εταίροι μας ε, και εμείς θα διαπραγματευτούμε την περαιτέρω μείωση του ελληνικού χρέους. Αλλά μην, ξεχνάμε όμως ότι η, συνεχής βελτίωση του λόγου χρέους προς, προς ΑΕΠ είναι η βελτίωση του παρονομαστή. Αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος και ο ασφαλέστερος τρόπος. Δηλαδή πρέπει, αυτό που πρέπει να πιέσουμε σήμερα είναι για περισσότερη ρευστότητα στην Ευρώπη για μια αποτελεσματική ε, ε τραπεζική ένωση, για καλύτερη χρηματοδότηση μέσω ίσω τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλων θεσμών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εμεί δεν κοιτάμε προ τα πίσω. Εμεί κοιτάζουμε, κοιτάζουμε μπροστά. Και, και, το μέλλον σαφώ είναι ευίωνο με βάση τι θυσίε του ελληνικού λαού, το τι έχουμε πετύχει μέχρι τώρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι έχουμε εξαλείψει ε, τα αίτια τη κρίση. Άρα Επιτρέψτε να σας πω ότι δεν συμμερίζομαι την απεσιοδοξία σας. Νομίζω ότι το μέλλον για την Ελλάδα και για, για, για τους Έλληνες είναι, είναι πολύ καλύτερο. Θα μου επιτρέψετε, ακόμα ε, ξέχασα να σας πω για τις τράπεζες, σαφώς πρέπει να υπάρχει ίση μεταχείριση, μεταξύ τραπεζών. Άρα εμείς διαπραγματευόμαστε σήμερα, ούτω ώστε οι όροι ε, που θα υπάρχουν για τις τράπεζες στην Ευρώπη να είναι παντού ίδια. Αυτό είπα το πρωί και στην, ε, και, και στην ε, και στα δύο κοινοβούλια, το ελληνικό και το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, όταν ερωτήθηκα, θα πρέπει οι όροι να είναι ίδιοι παντού. Όχι μόνο στην εγγύηση καταθέσεων, αλλά και στην κεφαλαιακή επάρκεια. Okay, e από την ε, ομάδα της Ευρώπης για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε, Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να συνεχίσω στο ίδιο θέμα το οποίο έφυξαν οι προηγούμενοι οδωρητές. Η Ελλάδα όντως, όντως έχει κάνει αλλαγές και μεγάλες αλλαγές, πρέπει να το δεχτούμε αυτό. Ωστόσο, το ε, τα ελλείμματα είναι μεγάλα και το δημόσιο χρέος είναι επίσης πάρα πολύ μεγάλο, φτάνει στα 180 δις. Και έχετε και πάρα πολλά δάνεια, τα οποία ε, καταλαβαίνουμε ότι βαραίνουν πάρα πολύ το ΑΕΠ σας. Η Ελλάδα επίσης θα πρέπει να επιστρέψει ε, τον επόμενο χρόνο 45,5 δις από το, τα δάνεια που έχει πάρει. Πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό. Εγώ είμαι από την Φιλανδία και η Πρωθυπουργό της Φιλανδίας ήδη έχει πει ότι η χώρα μας είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε κάποιες κινήσεις αλληλεγγύης προς την Ελλάδα. Χρειάζεστε περισσότερη αλληλεγγύη και από τις υπόλοιπες χώρες μέλη. Well, um, first of all, I want to make certain corrections to... Απάντηση. Να διορθώσουμε λίγο τα νούμερα. 320 και όχι 380, όπως είπατε, είναι το δημόσιο χρέος. και ενδεχομένως πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι ανακεφαλαιώσαμε τις τράπεζες. 40 δις δώσαμε λοιπόν για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Ε, αυτά λοιπόν είναι χρήματα τα οποία ε, θα ανακτηθούν αργότερα με την ιδιωτικοποίηση των τραπεζών στην Ελλάδα. Η κατάσταση λοιπόν είναι καλύτερη από όσο δείχνουν οι αριθμοί, εάν δει κανεί προσεκτικά και λεπτομερώς τους αριθμούς. Θέλουμε να μας βοηθήσουν οι εταίροι μόνο για να ξεκινήσουν οι συζητήσεις και οι διαπραγματεύσεις οι οποίες θα βασίζονται στις αποφάσεις του Eurogroup του Νοεμβρίου του 2012, δηλαδή για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει βιώσιμο το ελληνικό χρέος. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις, ας πούμε περαιτέρω μείωση του, των επιτοκίων, Επίσης ε, το να πληρωθεί, να γίνει η αποπληρωμή αργότερα, ε, χρήση του διαρθρωτικού ταμείου, αλλά μπορούν να υπάρξουν και άλλοι τρόποι. Θα πρέπει να είμαστε ετοιμοπόλεμοι και όταν ξεκινήσει η πραγματική συζήτηση σχετικά με την αηφορία του χρέους της Ελλάδος, να είμαστε έτοιμοι έτσι ώστε να βάλουμε στο τραπέζι καλές ε, ιδέες, ε, έτσι ώστε να γίνει βιώσιμο το χρέος και στην Ελλάδα και αυτό θα αποβεί και ε, σε καλό της Ελλάδας και των Ευρωπαίων εταίρων. Ευχαριστώ. Θέλεις να επανέλθεις? Όχι. Ο Χάντς Peter Μάρτι από τους μία εγγεγραμμένους τώρα. Ευχαριστώ. Μία ερώτηση μόνο υπό την ιδιότητά σας, του εκπροσώπου της Ελληνικής Προεδρίας. Ποια είναι η θέση σας για την επικείμενη μεταρρύθμιση των τραπεζών τη διαρθρωτική βάση της εκθέσεως Λίκανεν. Και η πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπής διαρκώς αναβάλλεται. Πώς το αξιολογείτε εσείς. Ουσιαστικά αυτό το καιρό περιμένουμε να κατατεθεί η έκθεση αυτή. Θα συζητηθεί προς το τέλος της Προεδρίας αν δεν απατώμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει τις προτάσεις της στα τέλη του μηνός και ε, εμείς θα το φέρουμε στο Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ. Έχω και άλλη ερώτηση. Εγώ δεν ρώτησα το διαδικαστικό, επί της ουσίας σας ρώτησα τη θέση σας παρακαλώ να μου πείτε, όχι τη διαδικασία. Μα δεν έχω δει ακόμα την έκθεση περιμένω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχω δει κάποιες εκθέσεις στον τύπο δημοσιεύματα, αλλά την ίδια την έκθεση δεν ε, την έχω υπόψη μου. Μα εγώ σας ρώτησα πολύ συγκεκριμένα, τα δημοσιεύματα είναι γνωστά. Η δική σας θέση ποια είναι από αυτόν. Uh, uh, my general proposition for, for... Η γενική μου πρόταση για τις τράπεζες ε, είναι ότι χρειαζόμαστε ένα υγιές τραπεζικό σύστημα ότι και ότι οι τράπεζες θα πρέπει να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να διασφαλιστεί αποφυγή ε, κινδύνων που αντιμετωπίσαμε ε, τώρα. Ξέρουμε τι συνέβη στο παρελθόν, έχουμε μάθει το μάθημά μας, ξέρουμε πώς προέκυψε η κρίση Ε, κατανοούμε πολύ καλύτερα ε, την κατάσταση ε, ξέρουμε γιατί διευρύνθηκε, διευρύνθηκαν τα ελλείμματα στον Νότο και γιατί έχουν, στον, στον Ευρωπαϊκό Νότο λέω, και πώς έχουν διονγκωθεί στον πλεονάσματα στον ε, Ευρωπαϊκό Βορρά. Τα γνωρίζουμε πλέον αυτά πολύ καλύτερα. Αλλά δεν μπορώ να πω τίποτα επί της ουσίας ε, πριν γίνει γνωστό. Αξιότιμε εκπρόσωπε του Συμβουλίου, πρέπει να σας πω το εξής. Αυτά που λέτε ε, δείχνουν τρομερή άγνοια των όσων θα κατατεθούν ως πρόταση. Ο λίκανεν ε, είναι η λέξη κλειδί και ο διαχωρισμός. Όταν βγαίνω στην ε, Αυστρία στο δρόμο και συζητώ με πολίτες εβδομάδες ολόκληρες, δεν βρήκα ποτέ πολίτη στο δρόμο που να έδειξε τέτοια άγνοια όπως αυτή που επιδεικνύεται εσείς αυτή τη στιγμή ταυτόχρονα σημαντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις λέγουν ότι το 90% των προβλημάτων των τραπεζών ε, δεν έχει λυθεί ακόμα και έχει μεγάλη σχέση με αυτή τη διαρθρωτική αλλαγή. Όταν έρχεστε στην Επιτροπή μας θα μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι θα έχετε διαβάσει, έχετε ακούσει τίποτα για την έκθεση Μακάρθη, από ό,τι φαίνεται όχι και να μην εκπλαγείτε που η ε, διάθεση απέναντι στην Ελλάδα, του κόσμου και τους πολιτικούς εκπροσώπους είναι αυτή που είναι. Και αν είστε τόσο επιτυχείς στη χώρα σας εσείς και επιδεικνύετε τώρα τέτοια ασχετοσύνη, πώς ερμηνεύεται αυτό το μεγάλο ρεύμα που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας και ενημερώνουν τους πολίτες σας πολύ πιο ε, καλύτερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια από ότι εσείς. Ως οικονομολόγος και πρώην τραπεζίτης μπορώ να απαντήσω πολλά, αλλά θέλω τώρα να μιλήσω ως πρόεδρος του ΕΚΟΦΗΝ, γι' αυτό πρέπει να προσέξω τι θα πω. Πρέπει να δω πρώτα την έκθεση της Κομισιόν πριν σχολιάσω. Μπορούμε να κάνουμε ανταλλαγή απόψεων για τον αμερικανικό τρόπο εδώ έχουμε μια έκθεση Μακάρθη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την ξέρετε. Αφήστε τον Υπουργό να απαντήσει παρακαλώ. Εδώ λοιπόν δεν είμαι ακαδημαϊκός θεωρητικός οικονομολόγος ή τραπεζίτης αλλά πρόεδρος του ΕΚΟΦΗΝ. Θέλω να δω πρώτα την έκθεση, την επίσημη έκθεση, όχι ότι διέρευσε στον τύπο, πριν να πούμε ότι θα μπορέσουμε να συζητήσουμε την έκθεση αυτή. Αλλιώς μπορούμε να κάνουμε χιλιάδες θεωρητικές συζητήσεις για το πώς θα διαχωρίσουμε τα είδη των τραπεζών πώς θα διευθετήσουμε τα εμπορικά, πώς θα υπάρχουν διαφορετικές ρήτρε για τις λιανικές τράπεζες και τις επενδυτικές κλπ. Αλλά αυτά είναι θεωρίες. Πρέπει να δω την έκθεση πριν κρίνω. Έχετε λίγη υπομονή. Uh, e και τώρα από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ο κύριος Λάγκεν. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κύριε Ποριέ, εδώ μπορεί ο καθένας να λέγει τη γνώμη του. Μην τα παίρνετε και όλα τις μετρητής αυτά που ακούτε, διότι ο συνάδελφος Μάρτιν εδώ δεν εκπροσωπεί σε καμία περίπτωση την πλειοψηφία μια πολύ μικρή ασήμαντη μειονότητα. Το λέω ειλικρινά. Ε, είναι θέμα ευγένεια ε, απέναντι σε έναν προεδρεύοντα υπουργό αυτό που πρέπει να δείχνουμε. Η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει τεράστιε προσπάθειε. Δεν χωράει καμία αμφιβολία περί αυτού. Και διαβάζω συστηματικά ελληνικέ εφημερίδε και διαπιστώνω ότι ε, τρέχουν στη δικαιοσύνη πολλές υποθέσεις για φοροδιαφυγή, ορισμένοι προκάτοχοί σας, μέλη κυβερνήσεων, βουλευτές, οι πάντες ε, έχουν ε, μπει σε ένα δρόμο τα πράγματα και είναι σωστός δρόμος για τις μεταρρυθμίσεις και το τονίζω και το υπογραμμίζω. Και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό που δεν έρχεστε εδώ να εξαγγείλετε τίποτα τεράστιες προγραμματικές δηλώσεις και τελικά ως προεδρεύον δεν μπορείτε να ξέρετε αν θα σας ακολουθήσει το Συμβούλιο. Το θεωρώ εξαιρετικό αυτό που λέτε, ότι αποφάσεις ακόμα και για τον μηχανισμό ε, SRM θα πρέπει να βασιστούν ε, σε μια ε, στιβαρή και γερή νομική βάση για τον νέο μηχανισμό εξυγίασης. Μην αφήσετε να σας τριμώξει κανένας. Αρκετή δουλειά έχει η Ελλάδα, πολύ σκληρός ο δρόμος και δύσκολος και εμεί θέλουμε να σας υποστηρίξουμε όσο μπορούμε. Αλλά αν επιμείνετε ότι οι αποφάσεις στο Συμβούλιο στη επιληθουανικής Προεδρίας όπως άκουσα από τη συνάδελφο Βόρτμαν Κον και την κυρία Φερέιρα, απλώς θα πρέπει να παραγωνιστούν παρόλα τα νομικά προβλήματα. Παρακαλώ να μην μπείτε σε αυτό το δρόμο, να μην υποκύψετε. Ε, παρακαλώ να βρείτε ένα δρόμο, αν γίνεται ένα συμβιβασμό και έτσι έχουν τα πράγματα. Ε, το άρθρο 114 ως νομική βάση για μια δεκαετία μέχρι να ιδρυθεί το Ταμείο αμφισβητείται. Αυτό δεν είναι καμία εφεύρεση κανενός ούτε του Συμβουλίου. Είναι γεγονός. Αν χρησιμοποιούνται ε, χρήματα από τους φορολογουμένους, από τους κρατικούς προπολογισμού, φορολογικά έσοδα για να δημιουργηθεί αυτό το Ταμείο υπάρχουν σε χώρες συνταγματικοί περιορισμοί. Και αν αυτό δεν το λάβουμε υπόψη δεν αυξάνεται η αξιοπιστία του Κοινοβουλίου ούτε μπορούν να αυτά τα πράγματα ε, υποπίεση. 1η Ιουλίου συνεδριάζει ε, για να συσταθεί σε σώμα το νέο κοινοβούλιο. Εάν δεν έχετε λύσει ε, το θέμα, η Τραπεζική Ένωση ε, δεν βιάζει και ελπίζω να μην δημιουργείται η εντύπωση ότι είναι τόσο πιεστικά τα πράγματα, γιατί δεν είναι. Well, thank you, Mr. Uh, σας ευχαριστώ κύριε Λάγκεν. Συμφωνώ απολύτως βέβαια με αυτά που είπατε. Μπορείτε να το φανταστείτε αυτό. Προσπαθώ να ακολουθώ τη λογική. Ξέρω ποια είναι η θέση του Κοινοβουλίου, ξέρω ποια είναι η θέση του Συμβουλίου. Έχω συμμετάσχει σε εργασίες. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι γίνεται καλύτερο και προσπαθούμε να ζήσουμε και σε, στον καλύτερο δυνατό κόσμο. Αλλά για να γίνει αυτό, όπως είπατε και, εσεί ο ίδιος, και εσείς ο ίδιος, πρέπει να έχουμε μια ισχυρή νομική βάση ε, έχει επιλεγεί μια βάση η οποία δεν είναι αρκετά σταθερή. Αυτό πρέπει να αποφευχθεί. Θα ήταν πάρα πολύ εύκολο να έρθω εδώ και να αρχίσω να σας λέω διάφορες ιδέες, αλλά δεν είναι ο σωστός τρόπος. Δεν πρέπει να ε, προχωρήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Θα πρέπει να έχουμε καλύτερη αμοιβαία κατανόηση, να συμμετέχουμε σε όλα. Θα έρθω εδώ οποτεδήποτε μου το ζητήσετε και θα σας αναφέρω ε, την πρόοδο κάθε φορά. Αλλά πρέπει να είμαστε όλοι υπομονετικοί, να είστε κι εσείς υπομονετικοί, να δείχνετε ευελιξία και σίγουρα δεν θέλουμε να παραγωνίσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τη διαδικασία. Ναι, βεβαίως μας ενδιαφέρει, λέει η Πρόεδρος, ε, και το περιεχόμενο, όχι νομική βάση. Από το ΕΛΚ, η Κορίν Βόρτμαν Κόλ. Ευχαριστώ. Εγώ αντικαθιστώ την κυρία Ντανούτα Χούμπνερ, την συνάδελφό μας από την Πολωνία και το ΕΛΚ που δεν μπόρεσε να προσέλθει. Έχει όμως μία ερώτηση για σας, θα τη διαβάσω. Εξετάζοντας τις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας για το ΕΚΟΦΗΝ, βλέπω ότι η διευκόλυνση για τη ισοζύγιο πληρωμών δεν εμφαίνεται, ενώ το θέμα είναι σημαντικό, καθώς η Προεδρία θα φροντίσει να καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις για τον ενιαίο μηχανισμό πληρωμών μπορεί να υπάρξουν όχι μόνο νομικά προβλήματα αλλά και πολύ σοβαρότερα. Εσείς βασίζεστε σε αυτά που μας είπατε ως προτεραιότητες αλλά δεν πρέπει να ξεχάσετε το σημαντικό αυτό θέμα της δημοσιονομικής και χρηματικής ε, βοήθειας και σε χώρες εκτός Ευρωζώνης. Η δημιουργία κάποιου καινούριου δημοσιονομικού εμποδίου στις χώρες αυτές θα ήταν αρνητική. Οι χώρες της Ευρωζώνης θα έχουν πρόσβαση τελικά στον μηχανισμό διάσωσης αλλά οι χώρες που δεν είναι στην Ευρωζώνη θα έχουν πρόσβαση μόνον σε έναν απαρχαιωμένο μηχανισμό η διευκόλυνση για το ισοζύγιο πληρωμών τους η Τραπεζική Ένωση δεν θα μπορέσει να καταλήξει ούτε στη Λιθουανική Προεδρία λόγω του ότι δεν συμφωνούν ακόμη πολλά κράτη. Κατά την Προεδρία σας, τι σκοπεύετε να κάνετε για να διευκολύνετε αυτή τη διαδικασία. Uh, we uh, Μελετούμε το θέμα αυτό. Νομίζω αν δεν σφάλω ότι χρειάζεται ομοφωνία στο Συμβούλιο το θέμα αυτό. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι προτεραιότητα, ωστόσο πρέπει να το συζητήσουμε και να δούμε εάν ε, ίσως ε, μπορεί να προωθηθεί η πολετονική προεδρία. So, Ναι. αλλά έτσι είναι δύσκολο με όλο, με την ε, ομοφωνία πραγματικά έχουμε πρόβλημα να επιτέχουμε. Ευχαριστώ πολύ, Σάρων. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Χαίρομαι. Χαίρομαι γιατί την επόμενη εβδομάδα θα σας έρθω στην Ελλάδα. Πολλά άλλαξαν από το πρώτο κούρεμα haircut. Τώρα έχουμε μια κεντρική τράπεζα η οποία έχει ε, το πρόγραμμα Draghi, ας πούμε, έτσι είναι γνωστό και γίνεται τελικά πιο αξιόπιστη ε, όσον αφορά τις αναδιαρθρώσεις ε, χρέους, γιατί αποφεύγεται η δυνατότητα επιμόλυνσης σαν αυτήν που είδαμε στην Πορτογαλία. Διάβασα στους Financial Times και ότι η κυρία Λαγκάρντα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ε, μάλλον φαίνεται να έχει προτείνει αναδιάρθρωση, νέα αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους και ότι επ' αυτού θα πρέπει να γίνουν διαπραγματεύσεις με τους άλλους πιστωτές, ε, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ε, καθώς επίσης και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στην ίδια εφημερίδα διαβάζω ότι φαίνεται ότι εσείς δεν το ζητήσατε αυτό στο Συμβούλιο γιατί φοβόσαστε αρνητική απάντηση του κ. Σόιμπλε. Καταλαβαίνετε ότι εμείς στην έκθεσή μας ζητούμε περισσότερο δημοκρατικό έλεγχο και της Τρόικα αλλά και των μελλοντικών ε, μηχανισμών βάσει της κοινοτικής ενωσιακής μεθόδου. Ερώτηση. Εάν υπήρχε αυτή αυτός ο δημοκρατικός έλεγχος. Εάν μπορούσε να υπάρξει περισσότερος δημοκρατικός έλεγχος όλων των μέσων αρρωγής προς τις χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα, θα ε, προσυπογράφατε μια τέτοια μέθοδο ε, και μάλιστα με την προϋπόθεση ότι μπορεί κάποια χώρα να το την πρότασή σας. Well, uh, Πρώτη ερώτηση. Ξέρετε ότι σε δύο Eurogroup συζητήσαμε το θέμα της χρηματοδότησης ε, του ελληνικού προγράμματος και επομένως ε, δεν είναι ότι κάποιος πρότεινε σε κάποιον κάτι άλλο και εγώ ήμουν μεσάζων ή οτιδήποτε. Ε, επιτύχαμε συμφωνία και είπαμε ότι υπό ορισμένε συνθήκες κάποια μέτρα θα έπρεπε να ληφθούν έτσι ώστε να μειωθεί έτσι περαιτέρω το ελληνικό χρέος. Επομένως δεν είναι ακριβές αυτό που μεταφέρεται. Έγινε ήδη συζήτηση στο Συμβούλιο επ' αυτού. Όσον αφορά τώρα την Τρόικα, γνωρίζετε ότι η Κομισιόν αναφέρεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, όσον αφορά τις ε, χώρες οι οποίες βρίσκονται σε συγκεκριμένα προγράμματα ε, και εγώ, εγώ πληροφορώ το Ελληνικό Κοινοβούλιο για την κατάσταση των πραγμάτων. Τώρα από εκεί και πέρα είμαστε ανοιχτοί για προτάσεις στο μέλλον μπορούν, μπορούν να βελτιωθούν τα πράγματα. Θα δούμε γιατί εμείς θέλουμε το καλύτερο για τις χώρες μας και για τους λαούς μας. Στην απάντησή μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασα ε, την άποψή μου σχετικά με το τι γίνεται στην Ελλάδα, σχετικά με την συνεργασία μας με την Τρόικα. Μπορείτε να διαβάσετε επακριβώς τις δηλώσεις μου στην απάντηση που έδωσα, που έστειλα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, έχω δηλώσει και ποια πήγαν καλύτερα, ποια πήγαν χειρότερα, ποια είναι ακριβώς η κατάσταση. Αλλά μερικές φορές νομίζω ότι απλώς θα πρέπει να μάθουμε από τα σφάλματά μας και το σημαντικό είναι με ποιο τρόπο μπορούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα στο μέλλον. Έχουμε μάθει από τα σφάλματά μας. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση του χρέους σε όλες τις χώρες που βρίσκονται σε πρόγραμμα, σε μνημόνιο ας πούμε και Νομίζω ότι ε, ε, βλέπουμε και στις τρέχουσες συναλλαγές ε, και στους, στο ισοζύγιο πληρωμών και στην, στα διορθωτικά βλέπουμε σε όλα τα στοιχεία να υπάρχει βελτίωση. Βεβαίως υπάρχουν και παιδεία επί των οποίων διαφωνούμε με την Τρόικα. Υπάρχουν μέτρα τα οποία υλοποιήθηκαν με καλύτερο τρόπο από ότι κάποια άλλα μέτρα. Υπάρχουν σημεία στα οποία βρισκόμαστε πιο πάνω πάνω από τους ε, στόχους. Ας πούμε, πετύχαμε πρωτογενές ε, πλεόνασμα μία, μία, ένα χρόνο πρωτύτερα. Ε, σε άλλες περιπτώσεις όμως είμαστε πάρα πολύ πίσω. Το σημαντικό είναι να βελτιώνουμε συνολικά την κατάσταση. Βεβαίως, τίνομαι πάντοτε ευήκονους στις προτάσεις σας. Βεβαίως, πάντα περιμένουμε και από εσά. Αλλά ε, ε, επαναλαμβάνω, η Κομισιόν αναφέρεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εμείς αναφερόμαστε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και οι άλλοι συνάδελφοι αντιστοίχω στα δικά του κοινοβούλια. Και νομίζω ότι ε, έχουμε ήδη δώσει αρκετέ λεπτομέρειε όσον αφορά την κατάσταση. Ευχαριστώ, αλλά μπορείτε να μας πείτε τίποτα παραπάνω για το τι έχει συζητηθεί στο Συμβούλιο ε, ε, ως προς το κούρεμα του ελληνικού χρέους στην αναδιάρθρωση. Δύο συνεδριάσεις της Ευρωζώνης καταλήξαμε, όπως είπα και πριν, ότι εάν η Ελλάδα πετύχει πρωτογενές πλεόνασμα και συνεχίσει η εφαρμογή των υπολείπων τμήματων του προγράμματος, τότε θα δούμε πώς μπορούμε να μειώσουμε περαιτέρω το ελληνικό χρέος και ως Έλληνας Υπουργός Οικονομικών απαντώ εδώ, όχι ως Πρόεδρος του Συμβουλίου. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, η κυρία Ροδικράτσα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, βλέπετε θα συνεχίσει η συζήτηση και στην Αθήνα και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό που μέλη της Επιτροπής μας με την ιδιότητα αυτή της σύνταξης της έκθεσης για την Τρόικα θα συνεχίσουν τη συζήτηση γιατί η ελληνική κατάσταση έχει πολλές παραμέτρους θετικές και πολλές προκλήσεις ακόμα και είναι πολύ σημαντικό να τις δουν επιτόπου οι συνάδελφοί μας και αυτά να αποτυπωθούν και στην έκθεση που συντάσσει η Επιτροπή μας. Ε, τώρα ερχόμενες δύο σύντομες ε, παρεμβάσεις με ερωτήσεις να κάνω κύριε Υπουργέ. Ε, είναι πολύ σημαντικό ότι εντάσσεται στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων την χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Δεν υποφέρει μόνο η χώρα μας, υποφέρει όλη η Ευρώπη, κυρίως ο Νότος και θέλω να σας ζητήσω να πραγματικά να θέσετε ψηλά στις προτεραιότητες στην ολοκλήρωση αυτών των δύο κανονισμών που ήδη θα ψηφιστούν άμεσα από την Επιτροπή μας για, τις, ε, για την εναλλακτική χρηματοδότηση. Ήθελα να ρωτήσω, ε, κύριε Υπουργέ, πώς πιστεύετε, ότι υπάρχουν ήδη εργαλεία στην Ευρώπη, αν δεν είναι ανεπτυγμένα όπως στις Ηνωμένε Παλιτείε, παραδείγματο χάρη, πώς περιμένετε αυτοί οι κανονισμοί με το πλαίσιο το, που δημιουργούν το ευρωπαϊκό θα, να βοηθήσουν τις προσπάθειες που γίνονται στις ε, διάφορες οικονομίες να έλξουν ε, χρηματοδότηση, τόσο για μακροπρόθεσμα έργα, όσο και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το άλλο θέμα, κύριε Υπουργέ, συζητήσαμε πολύ για το χρέος στην Ελλάδα. Είναι ένα πρόβλημα αναγνωρισμένο, εμείς το ζούμε έντονα σαν πιεστική πρόκληση στη χώρα μας, αλλά είναι και ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα, κύριε Υπουργέ. Ε, σαν προεδρεύον του ΕΚΟΦΗΝ έχετε κατά νου να εμβαθύνεται τη συζήτηση σε αυτό το θέμα της αντιμετώπισης του δημόσιου χρέους, διότι η Ευρώπη με όλο το ταλέντο και, το, και τη δυναμική που έχει βλέπουμε ότι δεν μπορεί να ανακάμψει εύκολα και ένα από τα θέματα, από το αβάρι της είναι το δημόσιο χρέος. Ε, έχετε κάποιες ιδέες ως εκοφήν. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κράτσα, ε, όσον αφορά το πρώτο, είναι ε, Πραγματικά η, απάντηση είναι ε, πολύ κρίσιμη. Κοιτάζουμε ε, τρόπους και πρακτικούς, κυρίως, για παράδειγμα, όπως ξέρετε, ε, στην Ελλάδα έχουμε χρησιμοποιήσει εναλλακτικούς τρόπους με εγκυοδοσία μέσω των διαθροτικών ε, μέσω των χρημάτων που παίρνουμε από τα διαρθωτικά ταμεία έχουμε προσπαθήσει μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζα Επενδύσεων να δώσουμε δάνεια και για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και, και για μεγάλα έργα. Αυτό είναι ένα πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Ε, επίσης ε, με συμμετοχή και ξένων κρατικών τραπεζών ε, δημιουργούμε ένα εργαλείο, το λέμε Institute for Growth, που θα συμμετάσχει, για παράδειγμα, και στο κεφάλαιο και θα δανειοδοτήσει επιχειρήσεις ε, ε, βιώσιμες, φέροντας ρευστότητα από το εξωτερικό και όχι παίρνοντας ρευστότητα από το ελληνικό σύστημα ε, και, και άλλες ιδέες. Κυρίως όμως προσπαθούμε να έχουμε ένα, ε, ένα ευσταθές τραπεζικό σύστημα, γιατί τελικά περί αυτού πρόκειται, αν δεν έχεις ένα, ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο στέκεται με σιγουριά στα πόδια του, τότε δεν θα υπάρχει εμπιστοσύνη. Αυτό λοιπόν προσπαθούμε να φτιάξουμε με την Τραπεζική Ένωση, ε, με όλα αυτά που κάνουμε για να έχουμε ένα ευσταθές τραπεζικό σύστημα στην Ευρώπη. Τώρα, στο ερώτημα ω προς το χρέος, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και παντού. όπω σα είπα και το, το, το πρωί, ο ασφαλέστερος τρόπο είναι να γυρίσει η Ευρώπη και κυρίως οι χώρες που έχουν πρόβλημα στην ανάπτυξη. Αυτό είναι ο πιο ασφαλής τρόπος για να μειωθεί το, το, το χρέος. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Ε, για παράδειγμα, αυτό θα έλεγα είναι ε, η απόλυτη προτεραιότητα. Σημαντικό ρόλο παίζουν οι αποκρατικοποιήσει. Η, η Ελλάδα, για παράδειγμα, είναι μια χώρα όπου ο δημόσιος τομέας έχει περιουσιακά στοιχεία αναλογικά με το ΑΕΠ περισσότερα από ό,τι έχει ο δημόσιο τομέα σε άλλε χώρε. Αυτό λοιπόν μα δίνει μια ευκαιρία μέσω αποκρατικοποιήσεων και να προσελκύσουμε ξένα κεφάλαια και να δημιουργήσουμε θέσει εργασία, αλλά και να μειωθεί περαιτέρω το, το ελληνικό χρέο. Από εκεί και πέρα όλε τι ιδέε που μπορεί να πέσουν στο, τραπέζι, έτσι, οι οποίε όμω ε, συμβάλλουν στην ευστάθεια και όχι στην αστάθεια του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, ε, συζητούμε. Ε, ναι, Now Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, κυρία Άννη Ποδηματά, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Σάρων. Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Θα ξεκινήσω από αυτή την τελευταία σας τοποθέτηση ότι ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του χρέους, όχι μόνο του ελληνικού συνολικά, είναι η ανάπτυξη. Αυτό προφανώς αφορά και στην περίπτωση του ελληνικού χρέους, της εξασφάλισης της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους. Ε, και θεωρώ ότι αυτή η διαρκώς ανακυκλούμενη ε, δημόσια συζήτηση περί περαιτέρω απομείωσης, κουρέματος, ε, είναι απολύτως επιζήμια και τελικά κουρεύει την αξιοπιστία της χώρας και άρα ε, δουλεύει σε βάρος της βιωσιμότητας του χρέους και νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει κάτι ώστε αυτή η δημόσια συζήτηση να πάρει τέλος. Για να έρθουμε όμως στην ανάπτυξη ε, που είναι ο ασφαλέστερος τρόπος για να εξυπηρετηθεί το χρέος, να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά του και να ε, πάμε στις πράξεις, γιατί μιλάμε για την ανάπτυξη και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, αλλά χωρίζει χάσμα αυτά που λέμε από αυτά που κάνουμε. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή είναι και στις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας, αν έχετε συγκεκριμένες σκέψεις, προτάσεις, έχει ψηφιστεί το Σύμφωνο Ανάπτυξης πριν από 1,5 χρόνο. Ε, συμφωνήθηκε από τους αρχηγούς κρατών έχει μείνει σε κάποια συρτάρια, δεν εφαρμόζεται. Σκέφτεστε να κάνετε κάτι για να το φέρετε ξανά στο προσκήνιο και να υλοποιηθεί. Δεύτερον, για την διαδικασία των Τρόικα, σας ρώτησε ο συνάδελφος Λίεμ, ε, εγώ θέλω να γίνω πιο συγκεκριμένη ως προς τους τρόπους ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας αυτής της διαδικασίας. Υπάρχει μια πρόταση που έχουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι και ψηφισμένη θέση, και αφορά στην ένταξη των χωρών που εφαρμόζουν πρόγραμμα προσαρμογής στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Όπως ξέρετε εξαιρούνται σήμερα οι τέσσερις χώρες που είναι σε πρόγραμμα. Ε, ούτως ώστε οι συστάσεις που περιλαμβάνονται στα προγράμματα προσαρμογής και ε, σε ό,τι αφορά το δημοσιονομικό σκέλος και σε ό,τι αφορά το διαρθρωτικό να εντάσσονται στη διαδικασία του εξαμήνου, στις συστάσεις αναχώρα, να συζητούνται ανοιχτά και να αξιολογούνται επιτρέποντας ε, επικαιροποιήσεις και διορθώσεις και στο πλαίσιο των προγραμμάτων. Θες ότι αυτή είναι μια πρόταση που αξίζει να ερευνηθεί, θέλω τη θέση σας. Και τρίτο και τελευταίο, είστε η πρώτη χώρα ε, μεταξύ των 11 χωρών που ανέλαβαν τη δέσμευση μέσω της ενισχυμένης συνεργασίας να εφαρμόσουν το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Ε, οι διαβουλεύσεις, οι διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο δεν πάνε γρήγορα και δεν πάνε και πολύ καλά. Το Κοινοβούλιο θέλει μια συμφωνία γρήγορα πριν τις ευρωεκλογέ. Θέλω να ρωτήσω κατά πόσο είστε διατεθειμένος να, ε, τρέξετε αυτή τη διαπραγμάτευση ώστε να έχουμε μια συμφωνία ε, πριν από τις ευρωεκλογέ του Μαΐου. Ευχαριστώ κυρία Ποδηματά. Θέσατε πολλά ερωτήματα. Θα προσπαθήσω να, τα απαντήσω. Ε, καταρχήν, να μιλήσουμε για ανάπτυξη για ανάπτυξη δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε εάν δεν λαμβάναμε μέτρα να ξαναφέρουμε τη χώρα στα πόδια της. Να αποκαταστήσουμε τη δημοσιονομική ισορροπία. Διότι ποια ανάπτυξη θα μπορούσαμε να είχαμε ε, με μια χώρα που είχε έλλειμμα πάνω από 10% του ΑΕΠ, που είχε πρω, πρωτογενέ έλλειμμα και στο προπολογισμό και στο ισοσύγιο τρε, τρέχουσών συναλλαγών. Άρα λοιπόν έχουμε αποκαταστήσει τώρα τι αναγκαίε συνθήκε για ανάπτυξη. Φυσικά αυτέ είναι μόνο αναγκαίε συνθήκε. Δεν είναι και επαρκεί. Ε, επαρκής θα γίνουν όταν πια αποκατασταθεί η ρευστότητα στην, στην ελληνική οικονομία και εκεί ε, τώρα είναι, είναι όλη μας η προσοχή. Ε, στο, επόμενο, στο αμέσως επόμενο διάστημα η ελληνική κυβέρνηση θα παρουσιάσει, ε, θα παρουσιάσει ένα σχέδιο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας για τα, για τα επόμενα δέκα χρόνια. Θα δείξει δηλαδή, κατά την άποψή της, πού θα πρέπει να είναι η ελληνική οικονομία 10 χρόνια από σήμερα, ε, τόσο από την πλευρά τη ζήτηση, όσο και από την πλευρά τη προσφορά, ποιοι είναι οι κλάδοι εκείνοι οι οποίοι αναμένονται να, να πρωταγωνιστήσουν και έτσι να δώσουμε στον κόσμο μια αίσθηση ότι α, οι θυσίε του ελληνικού λαού μέχρι τώρα πιάνουν τόπο και σε, και, σε ένα διάστημα από τώρα και στα επόμενα 10, 10 χρόνια θα έχει μια τελείω διαφορετική ελληνική οικονομία, ε, πολύ πιο ε, βιώσιμη, ε, με αναπτυξιακούς ρυθμούς υψηλότερους, ρεαλιστικού που θα στηρίζονται όχι πια σε κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα, αλλά σε εξωστρέφεια, σε καινοτομία σε εκπαιδευμένο και σε εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό είναι ο καλύτερο τρόπο να μειώσουμε και το χρέο. Διότι συμφωνώ μαζί σα ότι όλη αυτή η κουβέντα περί, περί κουρεμάτων και οι αιμονέ δεν κάνει καθόλου καλό. Ε, σα είπα πριν, το έχω πει σα σήμερα πέντε φορέ, ότι στο Eurogroup έχουμε συζητήσει και υπάρχει νομική βάση. Υπάρχει νομική βάση, όλοι συμφωνούν σε αυτό όταν έρθει ο χρόνος και ο χρόνος θα έρθει όταν συμφωνήσουμε με την Τρόικα στην τελευταία επισκόπηση ακριβώς θα δούμε πώς θα εφαρμόσουμε αυτή την απόφαση του Νοεμβρίου του 2012. Ε, Από εκεί και πέρα δεν έχω κάτι άλλο να πω πάνω, πάνω σε αυτό, αλλά συμφωνώ μαζί σας περί, περί της επιζήμιας ε, συζήτησης που, που, γίνεται, που, που γίνεται γι' αυτό. Ε, τώρα, για τη λογοδοσία ε, που είπατε και την ένταξη στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, συμφωνώ με τον Όλη Ρέν, είναι μια ενδιαφέρουσα πρόταση να, την εξετάσουμε. Σήμερα έχουμε ένα πλαίσιο στο οποίο, στο οποίο δουλεύουμε. Αν υπάρχουν ιδέε που θα βελτιώσουν αυτό το, το πλαίσιο, είμαστε όλοι αυτιά για να, ε, για να το συζητήσουμε. Ε, για το φόρο χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ε, μέσα από την ενισχυμένη συνεργασία των, των 11 χωρών προσπαθούμε να δούμε ποια είναι τα βασικά ζητήματα, ποια είναι η φορολογική βάση, ποια, θα είναι οι παράμετροι. Δεν έχει οριμάσει ακόμα. Όταν είναι όριμο θα έρθει στο ΕΚΟΦΗΝ για να το, για να το συζητήσουμε. Um, Σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν έχουμε χρόνο, όπως το είχα προβλέψει άλλωστε, για επιπλέον ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε που απαντήσατε στις ερωτήσεις και για τη χώρα σας, ενώ ε, ξέραμε ότι είπατε πολλά πράγματα που δεν αφορούσαν ακριβώς την Ευρώπη. Σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Προσβλέπουμε στην συνεργασία μαζί σας αυτό το δύσκολο θέμα του SRM ε, βεβαίως πρέπει να είμαστε υπομονικοί και ευέλικτοι, αλλά αυτό να μην ισχύει μόνο για μας, να ισχύει και για την πλευρά του Συμβουλίου. Βασιζόμαστε πάνω σας, ε, να ενθαρρύνετε τους συναδέλφους σας στο ΕΚΟΦΗΝ έτσι ώστε να πάρετε αποφάσεις προς τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. continue with Θα συνεχίσουμε ψηφοφορίες εντός ολίγων λεπτών. Μόλις καταλαγιάσει λίγο εδώ. Okay, Λοιπόν, πρέπει να συνεχίσουμε γιατί έχουμε ψηφοφορίες και τα καλά νέα είναι ότι θα ανεχτείτε και τις ανακοινώσεις της Προέδρου. Πρώτα απ' όλα λοιπόν μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι αύριο το απόγευμα δεν θα συνεδριάζουμε, μόνο πρωί. Παραμένει, διατηρείται το πρωί συνεδρίαση, αλλά η προγραμματισμένη για το απόγευμα ματαιώνεται. Δηλαδή θα τελειώσουμε το πρωί, θα προλάβουμε. Ε, αναθεωρημένο ε, χρονοδιάγραμμα για την έκθεση της Τρόικα. Επειδή η ad ε, ε, αποστολή αναβλήθηκε και συνδέεται με αυτό, έχουμε αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα και αυτό λέει ως εξής, προθεσμία κατάθεση τροπολογιών πλέον είναι Παρασκευή 31 Ιανουαρίου στις 5 το απόγευμα. Συζήτηση την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου εδώ των τροπολογιών θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ε, για να μεταφραστούν ως τότε. Αν θα είναι περιορισμένο το γλωσσικό καθεστώς, ελπίζω, ελπίζω να με συμπαθάτε. Ε, αν χρειαστεί θα συνεχίσουμε τη συζήτηση των τροπολογιών ε, ενδεχομένως την Πέμπτη στις 20 Φεβρουαρίου να μπει μια έξτρα περίοδος για να έχουμε στόχο να ψηφίσουμε στις 24 Φεβρουαρίου στην Επιτροπή μας στο Στρασβούργο και πάλι το απόγευμα. Ζητώ συγγνώμη γι' αυτό αλλά πρέπει να πάει το Μάρτι στην Ολομέλεια. Εμπιστεύομαι λοιπόν ότι μπορούν οι πολιτικές ομάδες να τηρήσουν αυτό το συμβιβασμό για το νέο χρονοδιάγραμμα και έχετε υπόψη ότι οποιαδήποτε αλλαγή διακυβεύει το στόχο και τις προθέσεις μας να πάει το Μάρτιο στην Ολομέλεια η έκθεση αυτή. Θα πρέπει όλοι να δείξουμε επικοδομητική στάση και πνεύμα συνεργασίας για να προκάνουμε. Ο οικονομικός διάλογος με την Ισπανία γνωρίζετε και θυμίζεται ότι πρόκειται να γίνει αυτό, θα ανταλλαγή απόψεων με τον Υπουργό Ντεγκρίντος που είναι ο, ο Υπουργός Οικονομικών της Ισπανίας την επόμενη Τρίτη 28 του μηνός στις 4 το απόγευμα. Επέφτει η μέρα πολιτικής ομάδας όμως αλλά έχει ζητηθεί και ε, διερμηνία για άλλες συνεδριάσεις, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε μικρότερο ρυθμό γλωσσών ε, από όσες χρειαζόμαστε σε αυτή τη συνεδρίαση. Ε, ζητώ και πάλι συγγνώμη, αλλά είναι σημαντικό να γίνει αυτή η συνεδρίαση με τον Ισπανό Υπουργό. Επίσης, μπορεί να χρειαστεί να ζητήσω συγγνώμη για να φύγω γιατί υπάρχει διακυβερνητική συνεδρίαση και πρέπει να είμαι εκεί. Ε, για τους τριμερείς διαλόγους, ενημέρωση. Ο πρώτος έγινε στις 16 Ιανουαρίου είναι για τις, ε, την οδηγία για τις πληρωμές. Γιούργεν Κλούτε ο συγητής μας, ε, για να υπάρχει μια ενιαία ορολογία και υποχρέωση να ε, υπάρχει ένας βασικός λογαριασμός για πληρωμές. Ε, το ξέρετε το θέμα έχουν ε, στις 11 και 26 Φεβρουαρίου δύο ημερομηνίες για διάλογο και το Μάρτιο θα προγραμματιστούν για να συμφωνηθεί πριν το τέλος της θητείας το θέμα σε πρώτη ανάγνωση. Επίσης μπορώ να σας πω για το τριμερή διάλογο για το SRM, ο δεύτερος έγινε στις 15 Ιανουαρίου για τον ενίο μηχανισμό εξυγίασης, η πρώτη ανταλλαγή απόψεων για τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων και ο καθορισμός της ε, σύνθεσης ε, του Διοικητικού Συμβουλίου και της διαδικασίας. Έχει δοθεί εντολή για τεχνικές ε, συνεδριάσεις ε, τέτοια θέματα εξυγίασης. Έχουμε κάπου συμφωνήσει και αυτό είναι ότι θα πρέπει να γίνει το συντομότερο Ε, να υπάρχουν κανόνες, ή κανόνες παιχνιδιού να γίνονται σεβαστοί. Ο επόμενος τριμερής διάλογος θα γίνει στις 29 συγγνώμη, Ιανουαρίου και μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν ε, διάφορα μέλη της διαπραγματικής ομάδας που θα παραμένουν στη συζήτηση για τη διακυβερνητική ε, συμφωνία. Έκαναν και κάποιες παρεμβάσεις. Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι συμφωνούμε με τη διακυβερνητική συμφωνία, αλλά καλό είναι να είσαι παρόν γιατί βοηθάει για τις διαπραγματεύσεις να ακούς τι διαμείβεται εκεί. Ε, και βεβαίως θα πρέπει να αποφασιστούν όλα γιατί δεν μπορεί κανείς να προχωρήσει σε ε, διακυβερνητική συμφωνία, αν δεν έχει συμφωνήσει να βγει κάτι από τη συναπόφαση. Αυτά θα τα ξαναπούμε για τα θέματα αυτά. Και τώρα μπορούμε να περάσουμε στις ψηφοφορίες. Τις κάρτες σας τις έχετε. Μπορούμε να ψηφίσουμε δοκιμαστικά για να δούμε πώς πάμε από κάρτες. Παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Δεν... Όχι, δεν άρχισε ακόμα. Δεν άρχισε. Α, έκλεισε κιόλα. Α, εντάξει, εντάξει, εντάξει. εντάξει. Μήπως είναι κανείς χωρίς κάρτα, ξέχασε την κάρτα του. Ο κύριος Γκερέρο. Ναι, ε, λίγα λεπτά θα διαρκέσει. Ε, αυτή τη στιγμή δεν έχω κάρτα, σε λίγο θα μου τη φέρουν. Αν υπάρξει κάποια ψηφοφορία που να αφισβητείτε θα σας πω πώς ψηφίζω, αν είναι πολύ μικρή διαφορά. Ωραία. Είναι καθοδόν η κάρτα σας, θα το δεχτούμε λοιπόν αυτό. Socialists, yes? I'm sorry, your group. I have no voting card okay. for a few minutes. Λέω ότι είναι καθοδόν η κάρτα μου, έχω στείλει να μου τη φέρουν. Εντάξει, εντάξει, θα το αντέξουμε. Okay. We've got Πέρας ψηφοφορίας 32 ευτυχείς ψήφισαν υπέρ, ένας δυστυχής κατά και 7 αποχές. We This is report. Ξεκινάμε λοιπόν. Με ποια έκθεση, με ποια, με ποια, ναι, Κούτας. this, this is the draft recommendation. So this is the short. Εδώ είναι η, ε, μικρή ψηφοφορία, αν θέλετε. Παράγραφος 1. Ίδια με την πρώτη παράγραφο ίντα. Σχετικά με τη συνένεση, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έχουμε την προφορική του εισηγητού για την παράγραφο 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έχουμε τεχνική ε, τροπολογία που δεν χρειάζεται να ψηφιστεί. Τώρα το τροποποιημένο κείμενο με ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ. Και θα προσθέσουμε και ε, μία ψήφο. Ψήφισαν όλοι να κλείσω την ψηφοφορία. 41 ψήφοι υπέρ, καμία ψήφιος ε, κατά, μία αποχή. Πολύ καλό αποτέλεσμα. Μπράβο. Ερχόμαστε τώρα στην, ε, στην έκθεση ε, Κούντα, ο πρόταση ψηφίσματος. Έχουμε αρχικό κείμενο πρώτη υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβασμός ε, A υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός B υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 6, κατά τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεν τα έκανα καλά. Δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 6, ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρας της ψηφοφορίας, 19 υπέρ 23 κατά, όντως έχετε δίκιο, απερίφθη. Είχα την αίσθηση ότι οι σοσιαλιστές ήταν υπέρ, αλλά κάτι δεν είχα υπολογίσει καλά. Τι να κάνουμε, σας καταλαβαίνουμε, σας καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, τροπολογία 7 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ, κατά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 κατά αποχές εγκρίνεται εκτιμώντας ένα μέχρι πέντε υπέρ κατά αποχές εν μπλοκ τις ψηφίσαμε Para 3A new there wasn't an original text there no okay that's fine I was just yes but it wasn't carried and there isn't any original text. So, so that was the amendment. Okay, just checking. Um, okay, now we'll do... Τώρα λοιπόν θα κάνουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία ε, το, την, ψηφο, την ψηφοφορία για το τελικό κείμενο. Άρχεται. Has everybody voted? One more to vote. Ψήφισαν όλοι. Votes closed and that is four. 40 ψήφοι υπέρ, καμία ψήφος κατά, τρεις αποχές. Μπράβο, μπράβο. Συγχαρητήρια. Εξαιρετικές επιδόσεις. Τώρα έχουμε την έκθεση του Βέρνερ Λάγκεν για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Βέρνερ. Ναι, μια σύντομη εισαγωγική παρατήρηση επιθυμώ να κάνω. Πρώτον, να ευχαριστήσω όλους τους συντονιστές και οδησιητές, καθώς επίσης και τις πολιτικές ομάδες που έχουμε βρει πολλούς συμβιβασμούς. Στο κεφάλαιο 7 θέλω να πω κάτι για τα ασφαλιστικά προϊόντα. Αναλογικά με τη συμφωνία για το MIFID πρέπει να ψηφίσουμε και πριν την Ολομέλεια να τα προσαρμόσουμε στον τριημερή διάλογο του MIFID για να υπάρχει συνέπεια και σαφήνεια της νομοθεσίας. Δεν έχουμε ακόμα τα κείμενα MIFID. Γι' αυτό θα ψηφίσουμε, αλλά το γράφει και το κείμενο σε μια αιτιολογική σκέψη, με την επιφύλαξη ότι θα προσαρμοστούν στα MIFID. Και παρακαλώ να ε, υπερψηφίσετε τους συμβιβασμούς και τελικά να δώσουμε διαπραγματευτική εντολή μετά τη λήψη απόφασης στην Ολομέλεια. Έτσι. Να μπει το MIFID 1 να συντονιστεί με αυτά που ε, θα προταθούν γιατί είναι τεχνικό το θέμα, δεν γνωρίζουμε σήμερα τι θα γίνει εκεί. Ωραία. Θα το δούμε αυτό όταν έρθει η ώρα του, αλλά το σημειώνουμε. Προχωρούμε. Συμβαστική πρόταση, α σε τρία τμήματα. Τμήμα πρώτο. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έχουμε ολίβι ρε παιδιά. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα υπέρ κατά ηλεκτρονικά καλύτερα ηλεκτρονικά είναι προφορική τροποποίηση του Σβέν Γκίγκολντ. Ηλεκτρονικά, ηλεκτρονικά. Ψήφισαν όλοι, μήπως λείπει κανείς, έληξε. Εγκρίνεται και το τμήμα 5 τώρα, περ, κατά, Ποχέ. πάλι ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Έληξε. Απορρίπτεται. Ωραία. Λοιπόν, τώρα πάμε στην τροπολογία 28. Στην επόμενη σελίδα. Λοιπόν, υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται νομίζω θα δούμε με ποια πλειοψηφία όμως ε, επαλήθευση για την 28 ψηφίσατε όλοι εγκρίνεται 24 υπέρ 18 κατά 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται με την ίδια πλειοψηφία συμβιβαστική β Υπάρχει πρώτα μία προφορική τροποποίηση για την αντικατάσταση της λέξης insured με τη λέξη customer. Υπέρ. Πρέπει να συνδυαστεί όμως με το τμήμα 1 μου λένε. Τμήμα 1 με τη λέξη insured αντικατεστημένη, αντικαθιστά τον customer. Υπέρ, κατά, αποχές, επανληθεύω επανληθεύω Ψήφισαν όλοι. Απορρίπτεται με μία ψήφο διαφορά. Τώρα πάμε στο τμήμα 1 χωρίς την προφορική τροποποίηση όπως είχε προηγουμένως δηλαδή υπέρ κατά εποχές Εγκρίνεται αυτό. Τμήμα 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τώρα συμβιβαστική γάμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 211 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 212 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 213 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 31 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση. Νομίζω εγκρίνεται αλλά επαλήθευση. Έλξη ψηφοφορία εγκρίνεται 24-19. Η 17 καταπίπτει, 215 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 7 υπέρ κατά α, ηλεκτρονικά, ηλεκτρονικά, ηλεκτρονικά. Ψήφισαν όλοι, έληξε. Εγκρίνεται 22-21. 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική δέλτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική σιγματάφ F δηλαδή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 225 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική ζήτα G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 228 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική τα H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική γιώτα προφορική τροποποίηση. Προφορική τροποποίηση. Με ή χωρίς την προφορική. Λοιπόν, συμβιβαστική γιώτα με την προφορική τροποποίηση υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Και τώρα χωρίς την προφορική τροποποίηση υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική J με την προφορική της τροποποίηση υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται ως είχε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ήμκο 12 καταπίπτει 241 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 242 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται όχι, ξανά θέλετε 242. Παλήθευση, εντάξει, εντάξει, παλήθευση. 242 ψήφισαν όλοι, έληξε, εγκρίνεται με τρεις ψήφους διαφορά. Ω, συγγνώμη. Τώρα, 243 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 245 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται αλλά θα επαληθεύσω. Η προηγούμενη είχε εγκριθεί αλλά όπως ξέρετε υπάρχουν και, διαφο και αλλαγές. Λοιπόν έληξε, εγκρίνεται με 5 ψήφους διαφορά. 244 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική κάπα πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική λάμδα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική μη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική νη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική όμικρον σε τέσσερα τμήματα. Τμήμα 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τμήμα 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τμήμα 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τμήμα 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα η 321 321 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 322 υπέρ κατά αποχές νομίζω εγκρίνεται επαλήθευσης Three more to vote, two more to vote. Τρεις ακόμη, δύο ακόμη. Ωραία, έληξε ψηφοφορία, εγκρίνεται 28 με 15. 324 υπέρ, κατά, ποχές, απορρίπτεται νομίζω. Θέλεις έλεγχος Βέν. λίγο κλείνει, κλείνει. Απορρίπτεται το ανάποδο δηλαδή. 323 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 325 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική π σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Νομίζω απέσχον οι σοσιαλιστές αλλά θα το παρελέξω, θα το ελέγξω. Θα ελέγξω. Έληξε εγκρίνεται με 10 ψήφους διαφορά. Τώρα η 340. 340 υπέρ. Κατά. Αποχές Επαλήθευση. Επαλήθευση. Έληξε. Απορρίπτεται. 341 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 342 υπέρ. Κατά. Αποχές Μερικοί περισσότεροι μου φάνηκε ψήφισαν υπέρ επαλήθευση. 342. 42. Απορρίπτεται με τρεις ψήφους διαφορά. 343 τώρα. Υπέρ κατά αποχές. Αποχές είπα. Επαλήθευση 343. Α, εντάξει, εγκρίνεται. Συμβιβαστική Q, υπέρ, κατά, ε. Α, όχι, όχι, τη ΣΥΜΚΟ έχει καταπέσει η 41. Λοιπόν, συμβιβαστική Q, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβιβαστική ρο, με την προφορική της τροποποίηση, υπέρ, κατά επαλήθευση της προφορικής τροποποίησης. Ε, επαλήθευση. Εγκρίνεται με 15 ψήφους διαφορά με την προφορική τροποποίηση. Συμβιβαστική σίγμα. Με άλλη προφορική τροποποίηση όμως πρώτα. Πρώτα ή με την προφορική. Υπέρ. Κατά α, τώρα δεν τα βλέπω καλά. Λοιπόν, με την προφορική τροποποίηση για τη συμβιβαστική S σε επαλήθευση. Επαλήθευση. Έληξε. Απορρίπτεται με 21 ψήφους διαφορά το αρχικό κείμενο της συμβιβαστική λοιπόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική ταφ. Στη σελίδα 31 την έχω λέει η πρόεδρος. Με η προφορική της τροποποίηση έχει αποσυρθεί. Λοιπόν, Συμβιβαστική ταφ ως είχε. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική ου. Με προφορική τροποποίηση. Υπέρ του τμήματος 1. Κατά αποχές επαλήθευση. Με συγχωρείτε, με παίρνει ο Ντράκη τηλέφωνο. Δεν μπορώ να σου απαντήσω, Μάριε. Close one, Έληξε. Εγκρίνεται με την προφορική τροποποίηση. Τώρα το τμήμα 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα συμβιβαστική Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική ωμέγα W υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική Χ σε ένα τμήμα αλλά καταρχήν με την προφορική της τροποποίηση υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται η αρχική χ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική α λάμδα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 625 Πω, μακριά είναι πολύ μακριά. Πολύ μακριά. 625 στη σελίδα 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Εβδομήντα τέσσερα υπέρ κατά χες απορρίπτεται. 626 υπέρ κατά χες απορρίπτεται. 96 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 627 υπέρ κατά χες επαλήθευση νομίζω απορρίπτεται 627 λοιπόν Απορρίφθηκε, απορρίφθηκε. 628 υπέρ. Κατά. Ποιες πάλι δεν κατάλαβα. 628 επαλήθευση. 628. Εγκρίνεται με τρεις ψήφους διαφορά. 657 εκπίπτει. Συμβιβαστική ΑΑ. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Ποιες Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά χες εγκρίνεται. Συμβιβαστική ΑΒ με προφορική τροποποίηση υπέρ κατά χες εγκρίνεται με την προφορική τροποποίηση. Συμβιβαστική ΑΓ πάλι με προφορική τροποποίηση υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται χωρίς την προφορική τροποποίηση λοιπόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται χωρίς Αλφα δέλτα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 656 υπέρ κατά Για να το επαληθεύσουμε. 656. Έληξε. Εγκρίνεται. 102 υπέρ. Κατά. Ποιες απορρίπτεται. Συμβιβαστική AG υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβιβαστική AH υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 662 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική AJ πρώτον με την πρώτη προφορική τροποποίηση Θέλεις να εξηγήσεις κάτι. Ναι, τέσσερις μήνες. Το είχε διορθώσει γραπτός ο συντάκτης της τροπολογίας. Έχει αλλάξει αυτό. Δεν έχει όπως γράφεται εδώ. Άρα δεν χρειάζεται να το ψηφίσουμε. Μάλιστα. Ψηφίζουμε 24 μήνες τότε μετά τη θέση σε ίσχυ. Ε, Κατά. Έχω μπερδευτεί τώρα. Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά και να μας εξηγήσει ο εισηγητής τι ακριβώς ψηφίσαμε εκ των υστέρων όμως. Α, είναι προφορική τροπολογία. Α, τώρα κατάλαβα. Ναι. Δεν πειράζει, εσείς πατάτε κουμπιά και βλέπουμε τι θα βγει. Τέσσερις δεν ψηφίζουν, ε. Δύο, ένας, μηδέν. Έλα, τελευταίος. Πάει. Πέρας. Μάλιστα. Απορρίπτεται γνησιότατο. Τώρα κατάλαβα γιατί το ψηφίσαμε. Λοιπόν, τώρα. Το αρχικό κείμενο που ήταν 18 μήνες. Έτσι δεν πρέπει να ψηφιστεί. Όχι. Συγγνώμη, ανοίγετε κανένα μικροφωνάκι να σας ακούμε. Αν κατάλαβα καλά, ψηφίσαμε πρώτα τους 24 μήνες και απερίφθη. Τώρα είναι το δεύτερο τμήμα και εδώ θα ήθελα να ψηφίσω υπέρ παρόλο που στον κατάλογο ψηφοφορία μας έχει αρνητικό πρόσημο. Προφορική του κυρίου Σβέν Γκίγκολτ, τμήμα δεύτερο. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο συντάκτη. Μα η, γραμματεία μου λέει πρέπει να ψηφίσουμε το αρχικό κείμενο για του 18 μήνε επίση. και μάλιστα πρώτα αυτό και μετά. Καλά, εμένα δεν με νοιάζει αυτό, λέει ο κύριο Λάγκεν. Είμαι υπέρ τη αναθεώρηση. Αυτό με ενδιαφέρει τώρα πότε θα γίνει. Ωραία. Πρώτα το 18 μήνο. Ψήφι υπέρ των 18 μηνών. Κατά. Αποχές. Πέρασαν οι 18 μήνες και όχι 24. Uh, και τώρα. Με την προφορική τροπολογία για την αναθεώρηση, ε, συμβιβαστική υπέρ, μαζί με την αναθεώρηση κατά αποχές εγκρίνεται αυτό. Και τώρα τελειώσαμε. Πάμε στην 106. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 107 υπέρ. Ορίστε. Όχι, όχι, πραγματικά πέρασε. 107 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 108 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 109 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 675 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 110 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 111 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 και λοιπές υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 113 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 114 έχει καταπέσει, 115 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 116 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τώρα με έχει συμπερδέψει. Ο εισηγητή απορρίπτει τι ίδιε τι τροπολογίε. Τι θα γίνει, να ελέγξουμε την 5. Να την ελέγξουμε. Γιατί πρέπει να καταλάβω τι γίνεται. Έλεγχο τη 5, παρακαλώ. Μα γι' αυτό τους έχουμε τους ελέγχους και τις επαληθεύσεις μεταξύ άλλων όταν κάποιος σφάλει. Ε, ψηφίσατε όλοι, Εγκρίνεται. Οι επόμενες καταπίπτουν και πάμε στην 119. Ψηφί Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 6 καταπίπτει και οι 2 επίσης. 120 ψηφί Τα τά αποχές απορρίπτεται. 121. Τμήμα πρώτον υπέρ. Κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 121. Ε, τμήμα πρώτον υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τμήμα δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 122 πρώτο τμήμα ψήφι κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Γιούρι 4 υπέρ έλεγχος για το δεύτερο τμήμα της 122 τμήμα δεύτερο ελέγχουμε. να ψηφίσατε όλοι. Εγκρίθηκε. 27-15. Γιούρι 4. Ψήφι Κατά αποχές εγκρίνεται. 1, 2, 3 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 124 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 125 υπέρ. Κατά αποχές ε, ε, απορρίπτεται. Η 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 127 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 8 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 131 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 133 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 136 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 134 τμήμα πρώτον ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές έλεγχος για το δεύτερο τμήμα παρακαλώ της 134 αρχίζει. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας εγκρίθηκε. Συνεχίζουμε. 135 τμήμα πρώτον. Ορίστε. Oh, έχουν καταπέσει αυτές οι δύο. Πάμε στην 138. Ψήφι Πέρα. Κατά αποχές εγκρίνεται. 10 ε, ψήφι πέρα κατά αποχές εγκρίνεται η συμβιβαστική αλφα μη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές μπορούμε να ελέγξουμε τη 12 παρακαλώ ηλεκτρονικά ψηφίσατε όλοι απορρίπτεται Άρα τώρα πάμε στην 154 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 153 υπέρ. Κατά αποχές. Νομίζω ότι έχει απορριφθεί, ας το ελέγξουμε όμως παρακαλώ. Άλλοι δύο να ψηφίσουν παρακαλώ. Πέρας. Ευχαριστώ. Α, εγκρίθηκε, μάλιστα. 155 είπε Κατά αποχές έλεγχος και για την 155. Ψήφισατε όλοι, εγκρίθηκε. 156 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 13. Ψήφι Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 157 σε δύο τμήματα. Α, όχι, έχει καταπέσει και τα δύο τμήματα. Οπότε θα πάμε μέσα στον 160. Ψήφι Κατά αποχές. Νομίζω ότι έχει εγκριθεί, αλλά στο ελέγξουμε για καλό και για κακό. 160. Έλεγχος. <laughs> Ψηφίσετε ακόμα δύο. Α, εγκρίθηκε. 14 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 161 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 162 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 164 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 165 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η επόμενη έχει καταπέσει 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 167 υπέρ. Όχι, όχι, αυτά καταπέσανε. Οπότε πάμε στα 170 υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. 171 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 172 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 173 υπέρ κατά αποχές ε, α, απορρίπτεται 174 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 175 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 176 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 178 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 179 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται καλύπτονται και οι επόμενες έτσι ε, συμβαστική αλφανή ναι, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 183 τμήμα πρώτον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές μπορούμε να ελέγξουμε παρακαλώ το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 183 Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίθηκε. 184 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 185 υπέρ κατά αποχές ας την ελέγξουμε παρακαλώ την 185 νομίζω ότι έχει απορριφθεί αλλά Συμφίσατε Ψηφίσατε όλοι. Απορρίπτεται. Άρα τώρα θα πάμε στην 186 είπε. κατά έλεγχος χρειάζεται και πάλι. Ψηφίσατε όλοι πέρας. Αγκρίθηκε. 23 καταπίπτει του εισηγητού. Ηλεκτρονικά το σύνολο του κειμένου ως τροποποιήθηκε. Παρακαλώ, αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Άλλος ένας. Κλείνει. Εγκρίνεται 35 υπέρ, 4 κατά και 3 αποχές. Το νομοθετικό ψήφισμα τώρα, ηλεκτρονικά επίσης. Ψηφίσατε όλοι. Συνεχίστε παρακαλώ. Άλλοι τέσσερις. Ένα κουμπάκι είναι. Πατήστε το σας παρακαλώ. Δύο. Πέρασε. Mm. Εντάξει, 43 τους έβγαλα. 37 υπέρ, 4 κατά, 2 εποχές. Ωραία. Τώρα, Βέρνερ, Λάγκεν. Τι γίνεται. Θα ήθελα να προτείνω να μην δώσουμε διαπραγματευτική εντολή, αλλά να το στείλουμε στην Ολομέλεια, ακριβώς λέγοντας ότι περιμένουμε τα κείμενα MIFID ε, και τα κείμενα του κεφαλαίου 7 θα πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτά για να μην υπάρχουν αντιφάσεις ε, και να συνάδει το κείμενο. Το έχουμε αποφασίσει άλλωστε και σε τροπολογίες αυτό. Ναι στην Ολομέλεια, όχι στη διαπραγματευτική εντολή. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ψηφίσουμε. Μάλλον όχι, δεν θα ψηφίσουμε. Εντάξει, ε, να το αφήσουμε στην Ολομέλεια. Νομίζω ότι θα πρέπει να το, όταν θα έχουμε τις αλλαγές MIFID να το αποσαφηνίσουμε. Ναι. Όχι, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Μπορεί να πάει στην Ολομέλεια. Ναι, ναι, Βέρνεν, πες μας, πες μας. Στη Μίφιτ υπάρχουν κάποιες μικρές αλλαγές που είναι πιθανές, πλην όμως όχι βέβαιες. Ο κανονισμός ΜΥΦΙΤ για τις ασφάλειες ε, μας έχει δώσει εμάς τη πιο σημαντική διαπραγματευτική εντολή. Ε, μπορεί να είναι μικρές αλλαγές που να μην χρειάζονται νέα εντολή. Ε, θα συμφωνήσουμε μεταξύ των σχεδόν εισηγητών της προσαρμογής και θα το στείλουμε στην Ολομέλεια. Όλα αυτά τα έχουμε συμφωνήσει. Ναι στην Ολομέλεια λοιπόν. Άρα ψηφίζουμε ότι θα πάει στην Ολομέλεια με τις τροπολογίες αν χρειαστεί και μετά θα αρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις μετά την Ολομέλεια. Ωραία. Υπέρ λοιπόν να πάει στην Ολομέλεια με όλα αυτά που είπαμε σχετικά με το MIFID και τις τροπολογίες. Θέλετε καλύτερη ηλεκτρονική ψηφοφορία. Όχι. Ναι. Ψηφίστε όλοι. Πρέπει να βρούμε την πλειοψηφία πρέπει να ψηφίσετε. Πέρας της ψηφοφορίας. Επομένως ψηφίσαμε 42 ψήφοι υπέρ. Καμία ψήφος κατά. Να πάμε στην Ολομέλεια με την, ε, τις αλλαγές της ΜΥΦΙΤ. Okay. Περνάμε τώρα στην έκθεση Wolf Klintz σχετικά με την μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Τελευταία ψηφοφορία είναι αυτή. Τροπολογία 13 υπέρ. Το ΕΛΚ να ψηφίσει παρακαλώ. Εάν θέλετε να απόσχετε, κανένα πρόβλημα. Αλλά πάντως, σας θυμίζω ότι ψηφίζουμε την έκθεση Κλίντς. Με παρακολουθείτε, λέει η Πρόεδρος. Έκθεση Κλίντς. Μακροπρόθεσμη χρηματοδότη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Αποχέσε. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο. Υπέρ. Αρχικό κείμενο. Υπέρ Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός A. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός α κεφαλαίο α μικρό. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 22 υπέρ κατά αποχές θα ήθελα να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 22. Πρέπει να ψηφίσουν δύο ακόμα συνάδελφοι και θα κλείσω την ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Κοιτάξτε, αν δεν σηκώνετε τα χέρια σας δεν βλέπω τα αποτελέσματα. Τροπολογία 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 24. Υπέρ κατά αποχές. Τι να σας πω, είναι δύσκολο. Για να κάνουμε μια ηλεκτρονική επαλήθευση. Right, closing the vote. Ψήφισαν όλοι πέρα στις ψηφοφορίες. And that's carried. 20... Εγκρίθηκε. Τροπολογία 25 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία, ε, τροπολογία 27 υπέρ. Κατά. Τι να σας πω. Ηλεκτρονική ε, επί της 27. Γιατί δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Τροπολογία 27. Two more to vote. Votes closing. Πέρας της And that's carried. Um, to the... Εγκρίνεται. Τροπολογία 28. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 29, 29 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τμήμα 2 υπέρ κατά Το τμήμα 2 παρακαλώ με ηλεκτρονική ψηφοφορία γιατί το ΕΛΚ δεν ξέρω πώς ψήφισε. Voted, votes closed. Πέρας της ψηφοφορίας. That's carried. Um, 35 in 35 υπέρ. Πάρα πολύ ωραίο. Κατά αποχές απερίφθη. 36 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 40 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 45 ηλεκτρονικός έλεγχος βεβαίως. Have you voted? Votes closed. Πέρας της ψηφοφορίας. Μάλλον τώρα θα κλείσω την ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 49 υπέρ. Κατά. να ελέγξουμε. Τροπολογία 49 ηλεκτρονικός έλεγχος. Um, can I open the vote, please? Close and open. Closing the vote. Votes closed. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 50 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 52 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 53 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται Εντάξει να ελέγξω λέει η Πρόεδρος αλλά το ΕΛΚ δεν σηκώνει τα χέρια του. Ένας ΕΛΚ σηκώνει και οι υπόλοιποι κάθονται. Πρόεδρε μετά από τόσα χρόνια δεν διαβάζετε πλέον με τηλεπάθεια τα αποτελέσματα. Δεν είναι δημοκρατικοί κανόνες αυτοί τέλος πάντων. Θα κλείσω την ψηφοφορία, παρότι οι δύο δεν έχουν ψηφίσει, εγκρίνεται. Δεν είμαι και σίγουρη τι ψηφίσαμε. Τέλο πάντων, το 53, ναι, το 53. Μπερδεύτηκα, λέει η Πρόεδρο. 55, υπέρ. Κατά. Mm Άποχε. Mm Ηλεκτρονική επαλήφωση για το 55. Τροπολογία 55. Άρχεται η λοιπόν. ψηφοφορία. Ηλεκτρονική. Όχι ηλεκτρονική. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, σας θυμίζω. Πέρας της ψηφοφορίας. Και εγκρίνεται. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 59 υπέρ. Κα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός B υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 76 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ψηφίζουμε την 78 υπέρ. Ε, Κατά αποχέσαι. απορρίπτεται 79. Όχι. Η ηλεκτρονική επαλήθευση για την 78. Παρακαλώ. I'm closing the vote. Vote's closed. Uh, and that's reject. Απερίφθη. 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 81 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 82 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός ΒΑ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 86 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Το πάμε στην 89 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός C υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μια προφορική τροπολογία στην παράγραφο 17α από τους σοσιαλιστές υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός Ή e και προφορική τροπολογία με την προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και πάμε τώρα στην 104 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, υπότιτλος 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 107 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 110 υπέρ. Ε, υπέρ 110 υπέρ κατά. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 110. πέρας της ψηφοφορίας και εγκρίνεται. 111 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 112 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 113 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβασμός ή e A υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 114 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 116 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 117 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, εν πάση περιπτώσει θα το δούμε μήπως άλλαξε το ΕΛΚ γνώμη 117 παρακαλώ 117. Δεν είμαι και σίγουρη ότι έχετε τον ίδιο κατάλογο ψηφοφορίας, εσείς οι δυο, εκεί. Μάλλον δεν είμαστε στην ίδια σελίδα. Πέρας της ψηφοφορία και απερίφθη. Τώρα πάμε στην τροπολογία 118. 118 υπέρ. Κατά αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 118, ωστόσο νομίζω ότι έχει απορριφθεί. Για να το δούμε. Ψήφισαν όλοι πέρας της ψηφοφορίας. Σας το είπα ότι είχε απορριφθεί. Έχουμε τώρα το αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 119 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 120 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, παράγραφος 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 123 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεν επισβήσουμε το αρχικό κείμενο. Τροπολογία 124 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 125 υπέρ κατά εκεί πίσω εσείς ψηφίζετε κατά εντάξει ηλεκτρονική επαλήθευση 125 γιατί μου λείπουν χέρια λέει η πρόεδρος Πόδια, Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 127 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 128 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία, τροπολογία 129 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβασμός G με προφορική τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται με την προφορική τροπολογία, αυτό ήθελε και το ΕΛΚΑ, να ελέγξουμε καλύτερα. Συμβιβασμός G με την προφορική τροπολογία των πρασίνων, εντάξει. εντάξει. πέρας της ψηφοφορίας και εγκρίνεται. 132 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 100 Η 132 δεν ψηφίζεται. <coughs> Τροπολογία 137 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός I υπέρ. Λοιπόν, ηλεκτρονικός έλεγχος ε, για το συμβιβασμό 1. Why didn't you vote γιατί δεν ψηφίσαμε την 133, θα, θα σας το πω μετά αυτό, αλλά να ολοκληρωθεί η ψηφοφορία για το συμβασμό I πρώτα. Λοιπόν, την 133 δεν την ψηφίσαμε γιατί ε, είχε, είχαμε περάσει την 132 και μετά η 133 ήταν συμβατή. Α, όχι, πρέπει να ψηφιστεί η 133. Ωραία, να ψηφιστεί η 133. Είναι η προηγούμενη σελίδα. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ωραία. 146 υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 147 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 150 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 28 υπέρ 149, άμα δεν έχω εγώ 149, τροπολογία 149 δεν έχω, λέει η Πρόεδρος. What number? I think 149 is included in some... some 149 has disappeared from my vote. Απολέστη 149. Κοιτάξτε, μετά την 150, έχω την 147, μετά έχω την 150 και μετά έχω την παράγραφο 28. Πού πήγε αυτή η απολεστήσα? Πού πήγε. Um, 149 Σας μιλώ εντύμως. 149 έχει εξαφανιστεί. Okay, it's gone into compromise AA. Α, μπήκε στη, στο συμβιβασμό α με κεφαλαίο α μικρό. Λοιπόν, παράγραφος 28 υπέρ. Κατά. Παρατηρήσεις εκτός μικροφώνου, οι διερμηνείς δεν ακούν. Ο Βέρνερ προφανώς δεν έχει την ίδια, τον ίδιο κατάλογο ψηφοφοριών, γιατί μου κάνει διάφορα σχόλια που δεν τα καταλαβαίνω. Και αυτή η τροπολογία στην οποία αναφέρθηκε είναι στο συμβιβασμό AA, α κεφαλαίο, α μικρό. Μάλλον έχεις ε, παλιά, παλιό κατάλογο, γι' αυτό μπερδευόμαστε. Συνεχίζουμε. Παράγραφος 28, αρχικό κείμενο, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έχουμε τώρα τα εκτιμώντας και τις αιτιολογικές. Από κοινού να τα κάνουμε on block, υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνονται. Και φτάνουμε στο συμβιβασμό J. Συμβιβασμός J. Έχετε δίκιο. Πρέπει να ψηφίσουμε πρώτα την αιτιολογική σκέψη A, υπέρ. Μπορούμε να ψηφίσουμε μέχρι το, το unblock μέχρι την 11α. Μετά την 11α τη θέλουμε χωριστά. Ωραία. Έχουμε το εκτιμώντας 11α, να το ψηφίσουμε χωριστά. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται παρόλα αυτά. Φτάνουμε τώρα την αιτιολογική σκέψη α, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβασμός J, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 4, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 7. Ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Έγκρινεται. Έχουμε τώρα την τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επανήλυψη για την τροπολογία 9 έχω αποχές που δεν μπορούσα να τις μετρήσω ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας και απορρίπτεται αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται προφορική τροπολογία στο, στην τελική σκέψη ΔΕΛΤΑ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, ε, γνωμοδοτήσεις ε, ε, καλύπτονται οι περισσότερες, ε, 4, ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, απασχόληση 9, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, απασχόληση 10, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και έχουμε και την 16 ε, της αποσχόλησης υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ρέτζι 12 υπέρ. Ρέτζι 12. Ε, Άσλι. Ε, εδώ στην τροπολογία 13 εγώ βλέπω ότι γράφει μέσα σε αγγίλες και ένα κείμενο. Είναι η employment 13. Εδώ λέει, στο, στη δικιά μου, στο δικό μου κατάλογο ψηφορές λέει ότι καλύπτεται. Εντάξει, θέλετε να το ψηφίσουμε. Παρ' όλα αυτά εμείς πιστεύουμε ότι καλύπτεται. Επομένως προχωράμε στην Ρέτζι 12, εκεί είχαμε φτάσει δηλαδή, Ρέτζι 12 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση για τη Ρέτζι 12. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Ρέτζι 13 υπέρ. Όχι, όχι, καλύπτεται. Άρα δεν ψηφίζουμε. Τροποποιημένο, ε, ψηφοφορία του τροποποιημένου κειμένου με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. 22 ψήφοι υπέρ, 2 ψήφοι κατά και 17 αποχές. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ όλους. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9.